meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer ersten Καλώς ήρθατε στην πρώτη συνεδρίασή μας της καινούργιας χρονιάς. Τις καλύτερες ευχές μου σε όλους σας από πλευράς Προέδρου και Γραμματείας. Κάποιους από εσάς ήδη σας είδα και είχα την ευκαιρία να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά και στους διερμηνείς, ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε και στα μέλη του προσωπικού που όλοι αυτοί μας βοηθούν να κάνουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, καλή χρονιά σε όλους, όλοι θα λάβατε το πρόγραμμα. Έχετε σχόλια, αν δεν έχετε σχόλια μπορούμε να προχωρήσουμε στο σημείο 1, την έγκριση της ημερήσιας ε, διάταξης. Υπάρχει και σημαντικό σημαντική αλλαγή. Η έκθεση για τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ενώσεω ε, θα αναβληθεί η συζήτηση, έτσι ζήτησε ο συγγητή. Ήταν σημείο 7 της ημερήσια. Λοιπόν, και θα ακολουθήσουμε τον Μάρτιο θα γίνει ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Αυτό που θα κάνουμε είναι το σημείο 15, το θέμα του κυρίου Κάλες, την έννοια του αποδεκτού κινδύνου. Θα το εξετάσουμε αυτό μετά την ακρόαση που θα έχουμε με τον Επίτροπο Φίντλ απόψε, σήμερα το απόγευμα μάλλον. Αυτά για, το, για την ημερήσια διάταξη, αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια. Σημείο 2, έγκριση των πρακτικών, συνηθισμένη διαδικασία εξετάστε το, το info της Κοκομπού όσον αφορά τα μέλη της Επιτροπής ο Χαν Ανρέ Ναράνχα Εσκομπάρ και ο Ντανιέλ Κασπάρη ο ένας αντικαθιστά τον άλλον εκ μέρους του ΕΛΚ εδώ μετά έχουμε το, τις εκπομπές μέσω διαδικτύου, το web streaming σήμερα και αύριο, αυτή η συνεδρίαση θα μεταδοθεί μέσω του web streaming στο διαδίκτυο, μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Και... Για συγχαρητήρια λένε ναι και από πλευράς Brown, Brian Gray, ένας ε, λογιστής και ελεγκτής και γενικός διευθυντής αναπληρωτής ε, παραμένει και γίνεται τώρα γενικός διευθυντής ε, ο Internal Audit Service, εσωτερική έλεγχη, οικονομική έλεγχη, συγχαρητήρια για αυτή την για αυτή την προβίβαση από την 1η Ιουνίου, έτσι, 1η Ιουνίου, σωστό, ωραία. Αλλά αποφασίστηκε ότι θα προβιβαστείτε. Και ταυτόχρονα αλλάζει ο εσωτερικός ελεγκτής Βάλτερ Ντεφά και παίρνει το αξίωμα Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης πάλι από την 1η Ιουνίου και εκείνος με αλληλομετάθεση. Αυτό ως γνωστοποίηση στοιχείων. Μπορούμε με αυτό να ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο στην ημερησία διάταξη. Ευχαριστώ. Περνάμε στο σημείο 4. Και πρόκειται για την χωρίση απαλλαγής για το 2007 το θέμα εκπαίδευσης, ε, κατάρτισης ε, πολιτισμού και νεολαίας αρμόδιος είναι ο Επίτροπος Γιάνν Φίγκερ. Ε, και δίνω όπως είχαμε προγραμματίσει τον λόγο πρώτα στον κύριο Λέβισον, μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεκτρικού Συνεδρίου. Θα λάβει πρώτο τον λόγο ο κύριος Λέβισον. Παρακαλώ, κύριε Λέβισον. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που παρουσιάζω το κεφάλαιο 9 του Ελεκτικού Συνεδρίου και την έκθεση για το οικονομικό του 2007. Το νέο κεφάλαιο 9 αφορά τον έλεγχο δαπανών, όσον αφορά την παιδεία και την ηθαγένεια και την ιδιότητα του πολίτου. Κάνουμε εισαγωγή. Κάνοντα την εισαγωγή στο κεφάλαιο 9, το, το ελεκτικό συνέθριο ήθελε να αντικατοπτρίσει την αλλαγή του προπολογισμού, διότι η πολιτική μα βασίζεται στι δραστηριότητε τώρα. Οι τομεί είναι στο κεφάλαιο 9. Εκπαίδευση και παιδεία, επικοινωνία, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη. Αυτά εντάσσονται εκεί τώρα συνολικά κονδύλια 1.188 εκατομμύρια ευρώ και 1.153 εκατομμύρια ευρώ. Ένα δισεκατομμύριο, εκατομμύρια δηλαδή. Είχαμε διαφορά από άλλα χρόνια λόγω της εισαγωγής νέων πολιετών προγραμμάτων και αυτό στα πλαίσια της περίοδου 2007-2013, του νέου δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτό συνοδεύτηκε από αλλαγή στο, στη δομή του εσωτερικού ελέγχου Μεγαλύτερη ευθύνη τώρα έχουν τα κράτη-μέλη. Απαιτείται οι εθνικοί φορείς να δίνουν ε, δελτίο αξιοπιστίας βάσει των δαπανών που γίνονται, λαμβάνουν χώρα στα κράτη-μέλη. Οι διαδικασίες του ελεκτικού συνεδρίου αποτελέθηκαν από δειγματοληψία 150 πληρωμών και από αξιολόγηση των συστημάτων ελέγχου και εποπτείας που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το δείγμα των 150 συναλλαγών κάλυψε 95 προκαταβολές και 55 ενδιάμεσες ή τελικές πληρωμές. Το ελεκτικό συνέδριο διαπίστωσε ότι 21% των πληρωμών επηρεαζόταν από ένα ή περισσότερα σφάλματα. Οι ενδιάμεσε και τελικές πληρωμές πλήττονται περισσότερο από σφάλματα από ότι προκαταβολές. Τα περισσότερα σφάλματα που διαπίστωσε το ελεκτικό συνέδριο αφορούσαν βασικά προβλήματα που αφορούσαν την επιλεξιμότητα των δαπανών και ανεπαρκή τεκμηρίωση των ε, αξιώσεων περί κόστος. Όσον αφορά την αξιολόγηση των συστημάτων ελέγχου και εποπτείας, το ελεκτικό συνέδριο έκανε μια αξιολόγηση σχετικά με το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφάρμοσε τον εισαχθέν σύστημα των εκ των προτέρων ε, δελτίων αξιοπιστίας όσον αφορά τους εθνικούς φορείς. Όταν κάνει την αξιολόγηση των δηλώσεων αυτών των δελτίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί ή να αποδεχτεί τις δηλώσεις αυτές αξιοπιστία και τους όρους ή να τα απορρίψει. Ε, εάν γίνει υπό όρους αποδοχή των δελτίων αυτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως να λάβει κάποια προληπτικά μέτρα. Όμως, ο έλεγχος των προγραμμάτων διαβίου εκμάθησης από πλευράς του ελεκτικού συνεδρίου έδειξαν ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα στις δηλώσεις εκ των προτέρων. Οι εθνικέ χρησιμοποιούσαν εθνικέ αρχέ διαφορετική βάση για τι εγγύησει και είχαν διαφορέ όσον αφορά την αποκάλυψη των διαδικασιών που πραγματοποιούσαν αυτέ οι αρχέ και αυτό οδηγούσε σε διαφορέ όσον αφορά την αξιοπιστία που διαπίστωνε όσον αφορά τι δηλώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια αξιολόγηση που περιοριζόταν σε μια εξέταση των συστημάτων και των ελέγχων θεωρητική, ενώ στην πράξη δεν έγινε παλίθε στα κράτη-μέλη πώ ακριβώς λειτουργούσαν οι διαδικασίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχθηκε όλε τι ε, δηλώσει ε, υπό ορισμένου όρους. Ο αριθμό των όρων που αφορούσαν του 39 φορεί ήταν 329 και επίκυλε από 3 μέχρι 13 όρου ανάφορα. Παρόλο που ε, κάποιου όρου αφορούσαν βασικά θέματα εσωτερικού ελέγχου όπω ομαδοποίηση των καθηκόντων, σύστημα εσωτερικού ελέγχου και ο τρόπος λειτουργίας των χρηματοστικών συστημάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν χρησιμοποίησε μέτρα προληπτικά. Επιπλέον, το ελεκτικό συνέδριο διαπίστωσε ότι δεν δόθηκε συνέχεια στι διαπιστώσει αυτέ, ούτε διευθυντικέ δράσει λομολογήθησαν, οι πολύ συχνά δεν ετηρήθησαν και 240 από του όρου που προποθέσει έπρεπε να εφαρμοστούν το τέλο του 2007. Και τέταρτον, μερικά από τα κριτήρια που χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της διαδικασίας αξιολόγησης δεν είχαν καθοριστεί επαρκώς και έτσι επικρατούσε μια βεβαιότητα όσον αφορά το τι σήμαινε η ολοκλήρωση της διαδικασία εξολογήσεως και ποια προληπτικά μέτρα θα μπορούσαν να αναλυθούν. Οι προαναφερθήσεις αδυναμίες μείωσαν την αξία των εκ των προτέρων δηλώσεων και της ειδικής διαδικασίας σαν στοιχείο του συστήματος ελέγχου και υποπτίας. Όμως, ο σχεδιασμός του συστήματος επίσης συμπεριλαμβάναν επισκέψεις ελέγχου στα κράτη-μέλη και αιτήσιες δηλώσεις εκ των υστέρων, δελτία αξιοπιστής των υστέρων. Το ελεκτικό συνέδριο θεωρεί ότι ένα τέτοιο σύστημα, αν εφαρμοστεί σωστά, θα μπορούσε να πετελέσει μια επαρκή βάση για να υπάρχει εμπιστοσύνη στο μέλλον. Ευχαριστώ. Όσον αφορά το δεύτερο Ευρωπαϊκό Ταμείο για το ελεκτικό συνέδριο έλεξε την προκαταρκτική αξιολόγηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Εθνικών Συστημάτων Εποπτεία και Έλεγχου. Τι έδειξε ο έλεγχο. Πρώτα απ' όλα ότι υπήρχαν κενά όσον αφορά τι περιγραφέ ε, των διαδικασιών ελέγχου και διαχείρισης που έδωσαν τα κράτη-μέλη. Η Δεύτερη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε διενεργήσει μόνο επισκέψει σε 10 κράτη-μέλη και περισσότερε επισκέψει δεν έγιναν εντό του χρονικού ορίου που έπρεπε εντό του 12 μήνου. Και τρίτον, η διαδικασία ελέγχου τη προόδου που πετέφει από τα κράτη-μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των διευθυντικών μέτρων θα έπρεπε να είναι πιο συστηματική. Στον τομέα των επικοινωνιών και των σχετικών δαπανών τη επικοινωνία, η έλεγχη εκ των προτέρων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι βασικό στοιχείο όσον αφορά το ελεγκτικό σύστημα. Το ελεγκτικό συνέδριο πίστωσε όμω ότι 7 από τα 12 σφάλματα που ενετόπισε θα έπρεπε να είχαν εντοπιστεί από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα α συνοψίσω ποια είναι τα συμπεράσματα του ελεκτικού συνεδρίου. Καταρχά, οι πληρωμέ που κατεβλήθησαν εντό του τομέα εκπαίδευση και ηθαγένεια επηρεάζονται από υλικά σφάλματα όσον αφορά την νομιμότητα και ε, τακτικέ πληρωμέ και αν υπάρχουν Αυτά τα σφάλματα λαμβάνουν χώρα διότι το νομικό πλαίσιο είναι περίπλοκο και τα κριτήρια επιλεξιμότητα είναι πολλέ φορέ ασαφή και πολλαπλά. Δεύτερον, εποπτική έλεγχη που διενεργούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Παιδεία και τον Πολιτισμό και σχετικέ δαπάνε και το, Ευρωπαϊκό, και το ERF2 είναι εν μέρει αποτελεσματικά. Το σύστημα, παραδείγματο χάρη για, τους, ε, ε, για την επικοινωνία, δεν είναι αποτελεσματικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βελτιώσει την αξιολόγηση των συστημάτων ρεποπτικών και ελέγχου που δημιουργούν τα κράτη-μέλη για το πρόγραμμα διαβίου εκπαίδευση και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για του Πρόσφυγε, αυξάνοντα τον αριθμό των επισκέψεων στα κράτη-μέλη. Και δεύτερον, θα πρέπει να βελτιώσουμε την πάροδο χρόνου την ποιότητα των εκ των ελέγχου που διενεργούνται ε, σε, με το σεβασμό των δαπανών για την επικοινωνία ελέγχοντας, έχοντας καταλόγους για σημεία πρέπει να ελέγχονται. Αν εφαρμόσει αυτές τις βελτιώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα οδηγούσαν οδηγίωση σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όσον αφορά τα ελεκτικά και βουλτικά συστήματα και για το πρόγραμμα διαβίου εκμάθησης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι σωστό δρόμο, τόσο ώστε θα βελτιώσει τη διαχείριση των δαπανών όσον αφορά την παιδεία και την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Λέβισον. Όπως είχαμε συμφωνήσει λοιπόν μετά από την εισαγωγή σας, ο Επίτροπος Φίγερ έχει τον λόγο παρακαλώ. Äh, ο κύριο Πρόεδρος, ο κύριο Μπός, ο κύριος, κύριε Σιγητά, κύριε Οντή, διακεκριμένα μέλη του Κοινοβουλίου και εγώ θα ήθελα να πω μερικά πράγματα απαντώντας τα εισαγωγικά σας λόγια και για τις ευχές που μας δώσατε για επιτυχία και, και εγώ εύχομαι να επιτυχές το 2009 να είναι καινοτόμο, έτος καινοτομίας και δημιουργικότητας. Έτσι το δηλώσαμε αυτό το έτος και πολλά ήδη ξεκίνησαν τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά αυτά τα ζητήματα πάνω σε αυτό το θέμα. Ο κύριος Λέβινσον στην, στα εισαγωγικά του σχόλια αναφέρθηκε συγκεκριμένα θέματα που αφορούσαν το, την έκθεση του 2007. Είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε στο Λουξεμβούργο πέρσι και θέλω να πω ότι πολλά ήδη εφαρμόζονται όσον αφορά τις συστάσεις αυτές. Το 2007 είναι έτος ουσιαστικών αλλαγών. Πρώτα απ' όλα είχαμε νέο νομικό πλαίσιο με προγράμματα νέας γενιάς για την περίοδο 2007-2013 και δεύτερον έχουμε εισαγάγει ένα νέο ελεγκτικό πλαίσιο για την εφαρμογή των λόγω προγραμμάτων όσον αφορά την, τα προγράμματα σε αυτό το τομέα ακολουθήσαμε τις συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου που ακούστηκαν και σε αυτή και σε προηγούμενες συνεδριάσεις και έχουμε συντονίσει καλύτερα τα προγράμματα και τις δράσεις τους. Χρησιμοποίησαμε πιο ομαδοποιημένα από όσον αφορά την χρηματοδότηση, ενίο έλεγχο, είναι πιο φιλικά για τους χρήστες τα προγράμματα, είναι πιο κοντά στους πολίτες, έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες κάθε χρόνο, μιλάμε για εκατομμύρια στον τομέα της υγείας ή στον τομέα του έρασμους ε, είναι πολύ δημοφιλή και σημαντικά προγράμματα για την Ευρώπη των λαών. Και σε αυτό το πλαίσιο του συστήματος ενιαίου ελέγχου έχουμε εισαγάγει εκ των προτέρων και εκ των υστέρων δηλώσεις όπως ανέφερε και ο κύριος Λέβινσον από την έποψη των κρατών μελών είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό και πιστεύουμε ότι αυτή η συνεργασία στον αφορά τον περιορισμό των ευθυνών είναι κάτι σημαντικό είναι νέα και συμπληρωματικά στοιχεία όσον αφορά την αρμόδια γενική διεύθυνση και το σύστημα ελέγχου. Αυτές οι συμπληρωματικέ δηλώσεις ενισχύουν έτσι περαιτέρω το ελεκτικό μας σύστημα που επιπλέον έχει διάφορα στοιχεία που βασίζονται στη διαδικασία. Λαμβάνονται υπόψη παλιές εμπειρίες τώρα όσον αφορά ε, έλεγχο συστήματων των εθνικών φορέων. Και τι συνέχεια δίνεται στις προτάσεις ε, επισκέψεις ελέγχου, συνεδριάσεις ενημερωτικές, κατευθυντήριες γραμμές κλπ. Η αξιολόγηση του ελεκτικού συνεδρίου όσον αφορά τα συστήματα ελέγχου και εποπτείας ε, τι διαπιστώνει λοιπόν το Εθνικό Συνέδριο, ήταν εν μέρει αποτελεσματικό το σύστημα, αλλά το όπω ακούσαμε, το Εθνικό Συνέδριο θεωρεί ότι ο σχεδιασμό του συστήματο, αν εφαρμοστεί σωστά, το σύστημα, αν εφαρμοστεί σωστά, μπορεί να δώσει επαρκή βάση για να υπάρχει βεβαιότητα και ασφάλεια στο μέλλον. Και αυτό είναι σημαντικότατο μήνυμα για τη συνεχή προσπάθεια που καταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση. Τρία, τρεις από τους τέσσερις τομείς ελέγχου που εξέτασε το ελεγκτικό συνεδρίο θεωρήθηκαν αποτελεσματικοί και είναι χρωματισμένοι πράσινοι τομείς. Έχουν σημειωθεί με πράσινη γραμμή. Η βασική εσωτερική έλεγχη είναι εκ των προτέρων έλεγχη των πληρωμών και εκ των υστέρων έλεγχη και εκ των υστέρων ε, αναλύσεις. Ο πιο σημαντικός τομέας που δεν θεωρείται αποτελεσματικός ήταν η αξιολόγηση των εκ προτέρων ε, δελτίων αξιοπιστίας που είναι νέα απέτηση που θα πρέπει να εφαρμόζεται στην έναρξη των προγραμμάτων. Λάβαμε υπόψη τις παρατηρήσεις του ελεκτικού συνεδρίου, πήραμε υπόψη πολύ σοβαρά και ήδη ε, ξεκίνησαν κάποιες δράσεις το 2008 ώστε να διορθωθούν αυτές οι αδυναμίες που ενετοπίστησαν στην αξιολόγηση των εκ των προτέρων δηλώσεων. Τέσσερα πράγματα θα ήθελα να αναφέρω διότι σχετίζονται άμεσα με τις συστάσεις όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο αξιοπιστίας όσον αφορά τους ελέγχους που διενεργούν οι εθνικοί φορείς όπως αποκαλούνται συνήθως τα Υπουργεία. Η Γενική Διεύθυνση για την Παιδεία και τον Πολιτισμό έχει εκδώσει συγκεκριμένε κατευθυντήριε γραμμέ για τι αιτήσει αυτέ δηλώσει και ήδη μάλιστα έχουμε διοργανώσει ειδικέ κοινέ συνεδριάσει με τι εθνικέ αρχέ τον Μάρτιο και τον Νοέμβριο πέρσι είχαν διοργανωθεί αυτέ το 2008 και οι επιτόπιε επισκέψει. Οργανώσαμε 33 τέτοιες επισκέψεις ελεγκτικές κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου έγιναν το τέλος του 2008 και κάλυψαν περίπου τους μισούς εθνικούς φορείς, οπότε έγιναν συγκεκριμένα πράγματα όσον αφορά τον άμεσο έλεγχο. Λοιπόν, λεχτή, οικονομικός έλεγχος. Στην ετήσιο έλεγχο του 2007 διενεργήθησαν αυτοί οι έλεγχοι και τα προγράμματα για υποπτικούς ελέγχους ήδη έχουν ξεκινήσει. Τρίτη απάντηση αφορά την, ε, τις διορθωτικές δράσεις και πώς παρακολουθούνται αυτές. Βασικοί έλεγχοι εντοπίζονται όπως αναφέρθηκε κατηγορίες ελέγχων και σύστημα βαθμονόμησης επίσης έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται για την αξιολόγηση των ετησίων αυτών δηλώσεων συμπεριλαμβανομένης και της συνέχεια που δίνεται στους όρους και προϋποθέσεις που δηλώνονται. Αλλά δεν υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις και όροι οι οποίοι να μπλοκάρουν τις διεργασίες μέχρι τώρα, μέχρι το τέλος του 2008 και αν προχωρήσουμε πολύ γρήγορα νομίζω ότι θα διεκπαιρωθεί το θέμα. Τέλος, ποια είναι η διασύνδεση μεταξύ βαθμολόγησης και των προληπτικών μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν. Το σύστημα βαθμολόγησης που έχει καταρτιστεί συσχετίζει σαφώς ένα βαθμό κάποιων χαρακτηριστικών με το προληπτικό μέτρο που θα πρέπει να αναλυφθεί. Δοθήσεις της έννοιας της πολιετούς εποπτικής στρατηγικής που ξεκίνησε το 2007, τη χρονιά που συζητάμε, και λαμβάνοντας υπόψη και τις δρομολογηθήσεις δράσεις βλέπουμε ότι τα εποπτικά και ελεκτικά συστήματα θα είναι πλήρως αποτελεσματικά από τη στιγμή που όλοι οι έλεγχοι και οι εποπτικές δράσεις έχουν εφαρμοστεί. Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά είμαι έτοιμος όχι μόνο να ανταλλάξω και άλλες απόψεις μαζί σας. Υπάρχουν πολλές απαντήσεις στο κείμενο και στις γραφικές παραστάσεις που έχουν επισυναθεί πρόσφατα αλλά θέλουμε να συνεργαστούμε περαιτέρω μαζί σας, με την Επιτροπή σας και με τον εισηγητή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Φίγερ. Περνάμε τώρα στη συζήτηση με τον Γενικό Εισηγητή που έχει τον λόγο. Παρακαλώ πια. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κρέη για τον διορισμό του, γιατί ο εσωτερικό έλεγχο είναι για μα πάρα πολύ σημαντικό και πραγματικά είναι σημαντικό που ένα άνθρωπο τόσο μεγάλη υψηλή ε, ποιοτική απόδοση ε, διορίστηκε σε αυτή τη θέση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίση την Κομισιόν που μα απάντησε καταρχήν γραπτά σε μια σειρά ερωτήσεων που είχαν υποβάλει οι ευρωβουλευτέ και ευχαριστώ επίσης για τις πρώτες προφορικές εξήγησεις. Και ήθελα επίσης να συγχαρώ το κρασμένο στο οποίο ανήκατε που πέρασε στην τάχτηκε στη ζώνη ευρώ. Και θα να σας πω ότι χαιρόμαστε που ξημερίσετε αυτό το περήφανο στοιχείο της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ για τις εξηγήσεις που μας δώσατε κύριε Πίτρο. Πέρα θα έχω να σας κάνω μια πρώτη ερώτηση που αφορά τον τρόπο της εφαρμογής γενικοποιημένα έμεσα και άμεσα. Γιατί ξέρετε ποιες είναι οι ευθύνε εκτέλεση από την Κομισιόν κεντρικά ή από τις εθνικές υπηρεσίες ή άμεσα από την Κομισιόν. Κατά τη γνώμη σας, ποιοι είναι οι λόγοι που αιτιολογούν τους διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης που ίσως για τους ε, πολίτες που εκπροσωπούμε φανούν ιδιαίτερα πολύπλοκοι. Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι τα πλεονεκτήματα των εθνικών υπηρεσιών σε σχέση με μια εκτελεστική υπηρεσία ή υπηρεσία διακανονισμού. Δεν ξέρω συνηθίζετε, κύριε Πρόεδρε, αλλά θα ήθελα να υποβάλω και στον κύριο Λεβίσον μια ερώτηση όσον αφορά τη μεθοδολογία ελέγχων του ηλεκτρικού συνεδρίου γιατί στο 9 φαίνεται ότι έχουν ε, αναλυθεί 150 ε, ε, συγγνώμη, φάκελοι. Αυτοί οι 150 φάκελοι θεωρεί το ηλεκτρικό συνέδριο ότι είναι αρκετοί σε σχέση με τον τεράστιο ρυθμό ε, συνολικών πληρωμών. Πόσες είναι όλες οι πληρωμές και 150 σαν δείγμα είναι επαρκές για να δημιουργηθεί μία άποψη βάσιμη και χωρίς φάλμα. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σοντή έδωσε μέρη την απάντηση νομίζω. Περίπλοκο είναι το σύστημα βέβαια. Ένα μέρο της περιπλοκότητας σε τι οφείλεται, στο ότι θέλουμε αυτά τα προγράμματά μας να πλησιάσουν τους πολίτες. Είπα ότι εκατοντάδες χιλιάδες είναι οι χρήστες των προγραμμάτων του τομέα της παιδείας ή της ηθαγένειας ή της νεολαίας και χαιρόμαστε διότι υπάρχει πολύ ισχυρή ε, ε, υποστήριξη πλευρά του Κοινοβουλίου. Κάνουμε περισσότερα ποιοτικά και ποσοτικά για να βελτιώσουμε την κινητικότητα που είναι, θα είναι η κινητικότητα έναν απόσπαστο κομμάτι της ε, εκπαίδευσης προετοιμασίας για μια καριέρα και την αριστεία. Το Εράσμους καλύπτει λιγότερο 4% των φοιτητών. Είναι μια μειοψηφία σε σχέση με τον πληθυσμό. Βασικός στόχος είναι να είμαστε κοντά στους χρήστες. Και δημιουργήθηκαν εθνικοί φορείς, κυρίως για τις δύο δράσεις. Για την παιδεία, το πρόγραμμα για τη διαβίου εκπαίδευση, το πρώην Σοκράτης, και δεύτερον είναι το πρόγραμμα για την νεολαία σε δράση. Σε περισσότερες χώρες είναι μία συν μία, συν, ένα συν ένας φορέας. Σε άλλες χώρες έχουμε περισσότερους φορείς. Έχουμε πάνω από 70 εθνικούς φορείς για αυτούς τους λόγους. Η συνεργασία μαζί τους είναι καλή, επικοδομητική. Συμφωνήσαμε ένα πλαίσιο ελέγχων και υπάρχει εμπιστοσύνη στα προγράμματα, αυξάνεται αυτή η εμπιστοσύνη. Είπα ότι υπάρχει μεγάλη υποστήριξη, γιατί είναι καλά προγράμματα και θεωρούνται ότι είναι ένα τμήμα τη πολιτική απαντήσεως των μέρων τη Ευρώπη. Αυτοί που ξέρουν την Ευρώπη μπορούν να ταυτιστούν με την Ευρώπη και πρέπει να δώσουμε στον κόσμο τη δυνατότητα να καταλάβει τα προγράμματά μας, τις πολιτικές μας και να συμμετάσχουν. Η αποδοτικότητα είναι υψηλότερη όσον αφορά την εφαρμογή μικρών υποτροφιών, μικρών δράσεων, όπου χιλιάδες επί χιλιάδων χρηστών χρησιμοποιούν διαδικασίες ρουτίνας για να υποβάλουν αιτήσει για να συμμετάσχουν Γι' αυτό αλλάξαμε κάπως δραστηριότητε και τι αναθέσαμε σε εθνικούς φορείς. Δημιουργήθηκε και ένας φορέας με, από κοινοτική θεσμική απόφαση μέτρα της Βρυξέλλες. Και αυτός ο φορέας βοηθά την υλοποίηση των δράσεων με αποκεντρωμένο τρόπο. Βοηθά αυτός ο φορέας να μειωθούν οι δαπάνες, βοηθά όπως είπα οι δράσεις να πλησιάσουν τον κόσμο διοργανώνει ενημέρωση, επικοινωνία, χρησιμοποιώντας τις γλώσσες των κρατών μελών. Υπάρχουν πολλαπλά ωφέλη που απορρέουν από αυτό το δίκτυο που αφορά τον τομέα της παιδείας και του πολιτισμού. Αυτά έχω να πω κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ακούσω και την απάντηση του συνεδρίου για τις πληρωμές. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι για μας αυτό το δείγμα των 150 συναλλαγών αρκεί. Τι κάνουμε. Κοιτάμε τις πληρωμές. Τις εξετάζουμε. Και γι' αυτό αρκούν τα 150 δείγματα. Πιστεύω ότι αυτό συνάδει και με τους διεθνείς ελεκτικούς κανόνες. Βέβαια, μπορεί να ακολουθήσει κανείς και διαφορετική δειγματοληψία. Σε κάποια γραπτά σχόλια του Επιτρόπου του κυρίου Φίγκελ αναφέρεται αυτό το θέμα. Και αναφέρονται και τα ερωτήματα του κυρίου Οντί, τα θέματα που έδειξε ο κύριος Οντί. Ίσως να υπάρχει και άλλος τρόπος. Νομίζω ότι ο τρόπος μας είναι σωστός όμως. Και έχω εμπιστοσύνη σε αυτό που λέω. Δεν ξέρω και ο Μπονίτσι ειδικό για τι δηλώσει αξιοπιστία και εισηγητή για τι δηλώσει αξιοπιστία έχει κάποια σχόλια πάνω σε αυτό. Ο κύριο Μπονίτς έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Βέβαια. Είναι πάντα καλύτερο να έχει κανείς μεγαλύτερο δείγμα. Όμως πιστεύουμε ότι το σφάλμα κυμαίνεται από το 2 με το 5% και έχουμε κάθε πεποίθηση ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Βάση του δείγματος. Έχουμε αναθεωρημένη προσέγγιση όταν παρά τις δηλώσεις αξιοπιστίας και τα απαραίτητα χέγγια. Είναι προσέγγιση που έχει αποδειχθεί. Θεωρείται λογική. Και κάθε χρόνο μας δίνει συνεπή αποτελέσματα. Από ό,τι γνωρίζω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διατείνεται ότι διαφωνεί με αυτή την προσέγγιση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από ό,τι άκουσα βελτιώνει, θέλει να βελτιώσει τα συστήματα για να πετύχει το ενδεδειγμένο επίπεδο αποτελεσμάτων. Με μικρότερα σφάλματα από αυτά που ήδη έχουμε εντοπίσει. Λιγότερα. Ναι, αν επιτρέπετε λέει ο κ. Επίτροπος, αυτό το θεώρησα σαν πρόσκληση να προσθέσω κάτι από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο ελεκτικό συνέδριο, στην έκθεση του συνεδρίου, βλέπουμε ποια εικόνα δημιουργείται, ποιο είναι το μήνυμα που διαβιβάζεται. Συγκρίνοντας τα στοιχεία, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό σφαλμάτων. Αυτό ο κύριος Λέβινσον και ο κύριος Μπονίτσι, συνάδελφοι του Λεκτικού Συνέδριου, περιέγραψαν. Ακόμα και σε αυτά τα ποσοστά ασφαλμάτων, με αυτά τα ποσοστά ασφαλμάτων, βλέπουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Άγκρη είναι, αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο κομμάτι το, της ευθύνης, πάνω από 80% των δαπανών. Αλλά τα σοβαρά σφάλματα είναι στο 13% στις άλλες δράσεις. 23% σε κάποιες δράσεις επικοινωνίας 29%. Τα Για τα περισσότερα χρήματα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι πιθανότητες σοβαρών σφαλμάτων ε, είναι πολύ χαμηλές. Και εστιαζόμαστε σε ευρύτερη αξιολόγηση πέραν των τελικών πληρωμών. Διότι εδώ μιλάμε για τελικές πληρωμές. Βλέποντας ποιο είναι το σημαντικότερο κομμάτι των δράσεών μας. Των δράσεων που οργανώνουν οι εθνικοί φορείς. Εκεί μπορούμε να πούμε ότι σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του 2007 που έχει δημοσιευτεί και είναι διαθέσιμη βέβαια, το ποσοστό των σφαλμάτων σε αυτό το τομέα είναι μικρότερο από 0,5%. 0,45% λέει η έκθεση για τους ελέγχους που διενεργούνται βάσει των συμφωνιών που καλύπτουν έμεσες κεντρικές δράσεις που ε, πραγματοποιούνται μέσω των εθνικών φορέων. Διαφέρει η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία και τα τελικά αποτελέσματα και το ποσοστό των σφαλμάτων ε, δείχνει το μέγιστο ποσό που αντιμετωπίζει προβλήματα. Χρήματα που μπορεί να ανακτηθούν και αν λαβούν υπόψη και άλλες πληρωμές, τα χρήματα που κινδυνεύουν, αν θέλετε, λόγω σφαλμάτων είναι πάρα πολύ λίγα, είναι χαμηλά τα ποσά, αυτό θέλω να πω. δεν είμαι σίγουρος αν συμφωνώ ότι αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσό τα μεγαλύτερα ποσά που κινδυνεύουν λόγω σφαλμάτων. Το πιθανότερο σφάλμα είναι μεταξύ, το ποσοστό είναι μεταξύ 2 και 5% το επίπεδο σφαλμάτων. Θα πρέπει να δούμε περισσότερα στοιχεία ότι αυτό είναι το μέγιστο ποσοστό σφαλμάτων. Α, αυτό είναι θετικό. Και τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί πράγματι κάποιες βελτιώσεις. Είναι θετικό αυτό. Είναι συνθετικό αυτό. Όμως δυστυχώς σε αυτή τη φάση Είμαστε μεταξύ 2 και 5%. Πόσες πληρωμές καταβάλλετε κύριε Επιτροπέ μέσα στα πλαίσια των αρμοδιότητων στο σύνολο. Πόσες. Uh, uh, Κοιτάξτε, τώρα οι απαντήσεις αυτές με αριθμητικά στοιχεία είναι ένα κομμάτι της γενικής απάντησης. Περίπου, περίπου μου λέτε λέει και ο Σοντή. 5 με 6 χιλιάδες. Αυτή είναι η απάντηση, λέει και ο Σφίγγελ. Όταν κοιτάξουμε την έκθεση του ηλεκτρικού συνεδρίου, έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχει ένα 21% σφάλματος αν το διαβάζω σωστά. Πράγμα που είναι τεράστιο ποσοστό. Ρωτάω λοιπόν, 150 δείγματα από πολλές χιλιάδες πληρωμών αρκούν για να εκτιμήσουμε το ποσοστό σφάλματος. Γιατί κατόπιν οι πολίτες διαβάζουν τις πληροφορίες αυτές. Και για μας μέσα στα πλαίσια της απαλλαγής που θα προετοιμάσουμε Πρόκειται για ένα τεχνικό θέμα ενδιαφέρον. Από ό,τι κατάλαβα, οπωσδήποτε θα είναι πάνω από το 2 ή από το 5%, αλλά πέρα από το ποσοστό σφάλματος, ο αριθμός των φακέλων που εξετάζονται θα πρέπει να μελετηθεί. 150 δεν μου φαίνεται ότι είναι επαρκή. Απάντηση σας ευχαριστώ πρόεδρο. Όπως είπα και όπως είπε και ο καθηγητής κ. Μπονίτσι, πιστεύουμε ότι είμαστε ε, σωστοί στο ποσοστό αυτό 2 με 5%. Μπορείτε να πείτε βέβαια ότι θα μπορούσαμε να το υπολογίσουμε στο μισό της εκατό αν θέλαμε, αλλά εμείς μπορούμε να σας αποδείξουμε τι κάνουμε ακριβώς. Και δύο τρίτα των δειγμάτων μας ήταν ε, προκαταρικές πληρωμές, ίσως στο μέλλον, αν πάρουμε προσωρινές και οριστικές συναλλαγές, ίσως πραγματικά το ποσοστό σφάλματος να αυξηθεί κάπως. Αλλά όπως ελεγχθεί θα πρέπει να δούμε και πόσα χρήματα θέλουμε να δαπανίσουμε για την εργασία αυτή στο ίδιο το ηλεκτρικό συνέδριο. Αλλά μπορούμε να είμαστε σχετικά ε, σίγουροι ότι περιγράψαμε πόσο, σφάλμα ήταν, πόσο υψηλό συγγνώμη, ήταν το σφάλμα και στους διάφορους τομείς και νομίζω ότι μπορούμε πραγματικά να υπεραμειθούμε των αποτελεσμάτων που έχουμε πετύχει εδώ γιατί είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε, συμμερίζομαι πολλές από τις ε, παρατηρήσεις του κυρίου Όντι, γιατί από τεχνική συζήτηση για τους αριθμούς καταλήγουμε σε πολιτικά μηνύματα και να υπάρχει μια διακμελοδοξία μικρή και να αντιμετωπίσουμε μεγάλη πιο ευρεία πραγματικότητα σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις εκτιμήσεις που γίνονται. όλα τα προβλήματα δεν μπορούσαν να καταμετρηθούν με τα σωστά ποσοστά ασφάλματος. Ο κύριος Λέβισον είπε ότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί και να συνεργαστούμε στενότερα και να ανταλλάξουμε τις ε, ιδέες μας για τη μεθοδολογία. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι απόλυτα έτοιμη να συνεργαστεί προσεχώς ακόμα και πιο στενά να μοιράζεται τις μεθόδους, τις εκτιμήσεις και για τα σφάλματα γίνει αξιοπιστία του συστήματος. Και τονίζω αυτό που είπε ο κ. Σόντι ότι είναι ένα σημαντικό μήνυμα προς τους πολίτες. Αυτό το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ κοντά προς τους πολίτες πιο κοντινό από οτιδήποτε άλλο θα έλεγα γιατί θα πρέπει να γνωρίζουν και να έχουν εμπιστοσύνη ότι αυτό το σύστημα είναι καλό, είναι για αυτούς, μπορεί να βελτιωθεί, θα πρέπει να βελτιωθεί και αυτή είναι η στόχη σε μια επταετή περίοδο, ιδίω σε επταετή περίοδο τη νέες γενιάς των προγραμμάτων. Αντί για συμφωνίες έχουμε βασικές αποφάσεις, πολύ πιο σύντομες περιόδους για τη λήψη αποφάσεων, μειωμένες προθεσμίες Πολλά θέματα έχουν βελτιωθεί στο σύστημα και έτσι τα προγράμματα θα είναι πιο ε, φιλικά προς τον χρήστη. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε και κύριε Λέβισον για τις απαντήσεις σας. Τώρα, όσον αφορά αυτό που σκεπτάσαστε για τα κράτη-μέλη. Είναι σημαντικό η Κομισιόν να έχει κάποια άποψη όσον αφορά την μοιρασμένη διαχείριση. Τι γνώμη έχετε για την εξέλιξη των πραγμάτων κύριε Επίτροπε, ιδίως όσον αφορά τις ε, δηλώσεις εξοπιστίας ε, ex ε, ante και ex post, εκ των προτένων και εκ των υστέρων Ποια είναι η απόψή σας για ε, τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη-μέλη για τα συστήματα αυτά ελέγχου. Έχετε την εντύπωση ότι το ποσοστό σφάλματος μειώνεται. Εάν ναι, θα μπορούσαμε εδώ να δώσουμε ένα καλό παράδειγμα στα κράτη-μέλη για να γενικοποιήσουν τις εθνικές αυτές δηλώσεις μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας απαλλαγής. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς πρέπει να πετύχουμε πιο στενή συνεργασία, επιμερισμό των ευθυνών όσον αφορά την αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών πολιτικών και προγραμμάτων. Θυμάμαι ότι όταν είχαμε αυτή την ιδέα υπήρχε κάποιος δισταγμός και σε κάποιες περιπτώσεις ε, έγιναν ε, ζωηρές συζητήσεις γιατί, κατά πόσο χρειάζεται, δεν θέλω τώρα να επιστρέψω στο τι έγινε πριν από δύο χρόνια, κυρίως το 2007. Πέρασε αυτό όμως, συμφωνήσαμε, όσον αφορά την αρχή. Μετά συμφωνήσαμε των λεπτομεριών, άρα υπάρχει ευελιξία του συστήματος, δεν υπάρχει ένα μοντέλο για τα πάντα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εσωτερική πρακτική ενός κράτους μέλους για τον έλεγχο. Εσωτερική έλεγχη, εξωτερική έλεγχη, διεξάγονται. Όλες οι χώρες όμως συνεργάζονται μαζί μας Συνεδριάσαμε δύο φορές πέρσι που σας είπα για να συμφωνήσουμε επί λεπτομερεστέρων ε, προσανατολισμών. Συναντηθήκαμε τον Μάρτιο και τον Νοέμβριο, άρα το σύστημα τώρα λειτουργεί. Επίσης υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι είναι υποφελές το σύστημα και συμπληρώνει αυτό το σύστημα την όλη φιλοσοφία που ακολουθούμε ή την πολιτική του ενιαίου ελέγχου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εποπτικός φορέας, τα κράτη-μέλη είναι στο επίπεδο του δευτερεύοντος ελέγχου και πρωταρχικό έλεγχος διεξάγεται επιτόπου από τους διάφορους φορείς. Δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν, έχει, δεν υπάρχει κάτι που θέλω να θίξω πάνω σε αυτό. Υπάρχουν αργές αντιδράσεις όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων ή των υστέρων δηλώσεις Τελικά παρελήφθησαν οι απαντήσεις και αυτή η αρχική περίοδος, η εισαγωγική περίοδος ε, δεν αποτέλεσε μόνο καλό μάθημα αλλά και σημαντική αλλαγή όσον αφορά την πολιτική και θεσμική προσέγγιση. Μοιραζόμαστε πολλά περισσότερα όσον αφορά την αξιοπιστία και την εκτέλεση των προγραμμάτων. Δεν θέλω να πω πολλά. Στο τέλος κάτι εξίσου σημαντικό αν συγκρίνω την προηγούμενη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την προηγούμενη πενταετία, ε, πρώτη με την τωρινή, είχαμε συνεργασία, πρόβλημα εκτέλεσης, τώρα έχουμε σαφέστερη συνεργασία, καλύτερη υποστήριξη όσον αφορά τους πόρους στην Επιτροπή Μπαρόσο και τον καθορισμό προτεραιοτήτων για τον προπολογισμό και καλύτερο επιμερισμό των ευθυνών όσον αφορά την ε, εκτέλεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο της κάθε χώρας, κάθε κράτους μέλους. Ο κ. Σοντή, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ε, εντάξει, καταλαβαίνω. Τα θετικά συναισθήματα όσον αφορά τον όλο μηχανισμό. Εξετάζοντας όμως τη θέση του ελεκτικού συνεδρίου, τι βλέπουμε. Ξέρουμε ότι είναι ένας φορές ανεξάρτητος το ελεκτικό συνέδριο και είναι πιο αυστηρό. Εξέτασε αυτές τις εκ των προτέρων δηλώσεις αξιοπιστίας και θεωρεί, θεωρεί ότι αυτές οι δηλώσεις ουσιαστικά δίνουν περιορισμένη δήλωση αξιοπιστία όσον αφορά τους ελέγχους. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα βαθμό μεγαλύτερο εμπιστοσύνη που δεν έχουμε. Τι πρέπει να γίνει κατά την άποψή σας συγκεκριμένα πράγματα έναντι των κρατών μελών. Και για αυτή την απαλλαγή το λέω, αλλά και για το μέλλον. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βλέπετε έχουμε επαφές με τα εθνικά κοινοβούλια και πρωταρχικός μας ρόλος είναι ο έλεγχος του, των διαφόρων ε, εκτελεστικών φορέων, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Εθνικά Κοινοβούλια Ελέγχου της Κυβερνήσης. Τι πιστεύετε, ποια στρατηγική μπορούμε να ακολουθήσουμε τόσο ώστε να λειτουργεί σωστά αυτό το σύστημα και να έχουμε υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνη και έτσι να μας δίνει θετική δήλωση αξιοπιστίας στο ελεκτικό συνέδριο απάντηση. Κύριε είναι μια διαδικασία. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να ξεκινήσουμε, έπρεπε να συμφωνήσουμε επί βασικών θεμάτων, όχι μόνο φιλοσοφικών, αλλά και πώς θα γίνει επιμερισμός των ευθυνών και πώς θα αναγνωρίζεται ο ρόλος καθενός. Το πετύχαμε αυτό. Ο πρώτος χρόνος ήταν μια αρχή. Ήδη κάναμε πολλά το δεύτερο έτος, όπως προανέφερα, σώσε το σύστημα να λειτουργεί ομαλότερα, αλλά λειτουργεί θα ήθελα να υπάρχει ένα τέτοιο επίπεδο εμπιστοσύνης ή συνεργασίας και σε άλλους τομείς πολιτικής όπου περισσότερα χρήματα χρησιμοποιούνται. Εμπιστοσύνη που θα υπάρχει στο μεταξύ του ευρωπαϊκού επίπεδου και εθνικού επίπεδου, π.χ. στα διεθνωτικά ταμεία, το χρειαζόμαστε αυτό για την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών δράσεων, των ευρωπαϊκών πολιτικών. Διότι συμφωνούμε επί των πολιτικών, των κονδυλίων και αυτά κάπου εκτελούνται στα κράτη-μέλη. Αυτό που επεξεργαζόμαστε τώρα είναι εκ των υστέρων δηλώσεις. Κάναμε κάποια πράγματα και η κυρία Γενική Διευθύντρια έστειλε κάποιες επιστολές στα κράτη-μέλη όπου εκεί ζητούμε να είναι προσεκτικά τα κράτη-μέλη να στέλνουν απαντήσει έγκαιρα. Όλες οι απαντήσεις είναι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα γίνει πλήρης αξιολόγηση συντομότατα και νομίζω ότι για τις μελλοντικέ εκθέσεις τα επόμενα χρόνια μπορούμε να αναμένουμε πραγματικές βελτιώσεις. Προσωπικά είμαι ικανοποιημένος που το πρώτο έτος απετέλεσε μια αρχή και όλες χώρες χωρίς να υπάρχουν σημαντικές διαρρέσεις μπόρεσαν να δουν τη σημασία της προσπάθειας και να συμφωνήσουν επί των αρχών που εφαρμόζουμε, επί των προσανατολισμών των κατευθυντηρίων γραμμών που συμφωνήσαμε και εφαρμόζουμε εντό του συστήματο. πολιτικός είναι προαπαιτούμενο αυτό. Συμφωνώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι εν γέννη ήδη έχουμε πει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την παρέμβασή μου και από την έκθεση, έχουμε πει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι καλά τα πάει, σωστό δρόμο ακολουθεί, όλοι πρέπει να εφαρμόσει και τις συστάσεις μας και ακούμε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπόσχεται να συμμορφωθεί και ήδη έκανε πολλά και είμαι πολύ χαρούμενος που τα ακούω αυτά. Βεβαίως το ελεγκτικό συνέδριο αποτελείται κυρίως από ελεγκτές και πρέπει να κάνουμε ελέγχους και μετά θα επανέλθουμε το επόμενο φθινόπωρο για να δούμε πώς πήγαν τα πράγματα. Εγώ ελπίζω ότι πήγαν καλά τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα οι ετήσιες δηλώσεις ε, αξιοπιστίας ε, για το 2007 θα έπρεπε να έχουν υποβληθεί ε, από τα κράτη μέχρι τον Απρίλιο του 2008. Αυτά θα έχουν πιστεύετε επιπτώσεις στις δηλώσεις τάση για το 2008. we got, most of them in time. Κοιτάξτε, πήραμε τις περισσότερες απαντήσεις γέρος. κάποιες καθυστέρησαν. Ε, ζητήσαμε προσοχή και συνέπεια διεκπεραιώνονται υποθέσεις και το τέλος του μήνα θα είμαστε έτοιμοι θα έχουμε και τα 27 κομμάτια του μοσαϊκού, σχηματιστή εικόνα. Έχει, ε, δημιουργήθηκε μια ορμή το 2007 όσον αφορά τη οργάνωση των νέων προγραμμάτων και του συστήματος. Χρειάζονται και άλλες βελτιώσεις η κατάσταση δεν είναι ίδια σε όλα τα κράτη. Είπαμε, είναι μια εικόνα αποτελείται από κομμάτια, ένα μοσαϊκό, ένα ψηφιδωτό και δεν υπάρχει κάποια προβληματική χώρα ή κάποιος προβληματικός φορέας που θα πρέπει να αναφέρουμε και να λάβουμε μέτρα. Είπαμε ότι πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις θα μπορούσαν να ληφθούν κάποιε αποφάσει γιατί κάποιε φορέ τα πήγε καλά ή παρέψε κάποια πράγματα. Δεν χρειάστηκε. Αυτή είναι μια απάντηση. Άλλη απάντηση. Πιστεύω ότι με την κοινή αυτή προσέγγιση και το ενίο σύστημα ελέγχου βελτιώνουμε τα πράγματα περαιτέρω και αν επικοινωνεί ενεργά το ελεκτικό συνέδριο πάνω σε αυτά τα θέματα, στα πλαίσια της ανεξαρτησίας του, μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα πιο γρήγορα το σύστημα. Αυτά. Ευχαριστώ κύριε Πέτροπε. Θα μπορούσατε να μας πείτε με δύο λόγια τι πιστεύετε για την απόσταση που πιστεύουν υπάρχει μεταξύ του εθνικού της εθνικής έκθεσης ε, την εξήσεξη και της άποψης του λεκτικού συνεδρίου. Mm. Maybe uh, Ίσως η Γενική Διευθύντρια θα ήθελε να προσθέσει κάτι εδώ σχετικά. Το θέμα ένα ερωτηματικό δηλαδή αν θα ήταν εύθετο να υπάρξει κάποια επιφύλαξη για την έκθεση ή για την εφαρμογή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2007. Πιστεύω ότι είχαμε δίκιο και είχε δίκιο και η κυρία να μην το κάνουμε αυτό. Και η ίδια η πρακτική έδειξε ότι ήταν ορθή αυτή η ανοιχτή προσέγγιση. Αφενός υπάρχουν κίνδυνοι και προβλήματα. Από την άλλη πλευρά υπήρξαν βελτιώσεις. Κάναμε πολλά πρακτικά πράγματα ως ε, πρακτικά βήματα προς την ορθή κατεύθυνση που υιοθετήσαμε. Όλες αυτές οι αδυναμίες λοιπόν δεν ε, οδήγησαν σε μια υποχρέωση να υπάρξει κάποια επιφύλαξη, αλλά για τον προβληματισμό σχετικά που δεν οδήγησε στην ε, επιφύλαξη. Πιστεύουμε απόλυτα ότι ήταν πολιτικά ορθή κίνηση. Επίσης και σε σχέση και με την ε, συνολική επιβράδυνση ή καθυστέρηση προγραμμάτων που αφορούν τους ε, πολίτες και φυσικά υπήρχαν και άλλοι κίνδυνοι που ε, θα συνεπαγόντουσαν αν υπήρχε καθυστέρηση έναντι των εθνικών αρχών και φορέων για πάρα πολλούς που εμπλέκονται δηλαδή στην πρακτική σε αυτά και η γενική αξιολόγηση συνολικά έδειξε ότι ήταν ορθή αυτή η αποτίμησή μας. Επιβεβαιώνω και παληθεύω λοιπόν ότι ήταν ορθή αυτή η προσέγγιση αυτή που υιοθετήθηκε και τα συνολικά αποτελέσματα επαληθεύουν, επιβεβαιώνουν αυτή την ορθότητα, την ε, θα έλεγα το λελογισμένο ή την σοβαρότητα της θέσης ε, που υιοθέτησε η Γενική Διεύθυνση. Ευχαριστώ. Uh, uh, να σας υπενθυμίσω ότι προβλέπεται κάποιος από τους υπαλλήλους να μπορεί να παρέμβει αν θεωρεί ότι πρέπει και ότι αυτό είναι εύθετο. Η κυρία Κοκτάν παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μία διευκρίνηση ήθελα να κάνω τα δύο περισμένα έτη είχαμε μια επιφύλαξη για το θέμα των εθνικών υπηρεσιών. Δεν το έκανα το 2007 για τους λόγους που εξήγησε και τους Επίτροπος. Και γιατί το 2007 και το επιβέωσε το ηλεκτρικό συνέδριο, λέγοντα ότι η βάση του συστήματος είναι καλή, με λέω ένα σύστημα που μας επιτρέπει να μην ε, έχουμε μια επιφύλαξη γιατί μπορούσαμε να έχουμε επαρκείς διαβεβαιώσεις. Εκεί που κάνει κάποιες επιφυλάξεις στο ηλεκτρικό συνέδριο είναι η εφαρμογή του συστήματος του 2007. Εγώ θεώρησα ότι η αρχή ήταν η λογική. Το 2007 το εφαρμόσαμε σταδιακά, το βελτιώνουμε το 2008 όπως ανέφερε και ο κύριος Επίτροπος και αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη ακόμα εμπιστοσύνη από ότι ε, στο παρελθόν. Μπορώ τώρα να είμαι αρκετά σίγουρη. Η διαφορά είναι το 2007 η εφαρμογή του σήματο επέτρεπε να κάνει το καλό. Εγώ πιστεύω ότι πρόκειται για ένα σύστημα που εισήχθη για να έχουμε κάποιες λακές διαβεβαιώσεις. Ο, ο κύριος ε, ε, Λεβίσον είπε ότι πρόκειται για τη σωστή βάση. Και εγώ βασίστηκα στο σύστημα που είχε εισαχθεί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Euh, Ευχαριστώ κύριε Γενική Διευθύντρια. Κύριε Επίτροπε, μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια όσον αφορά τα πραγματικά πλεονεκτήματα της εκτελεστικής υπηρεσίας που δημιούργησε η Κομισιόν σε σχέση και με το παλαιό σύστημα, δηλαδή τα γραφεία αυτά ε, τεχνικής ενίσχυσης. Το προηγούμενο σύστημα ανήκει στην ιστορία με πολλά ερωτηματικά λόγω δυναμίων. Η δημιουργία του εκτελεστικού φορέα αυτού για θέματα οπτικοκουστικά παιδείας και πολιτισμικά θέματα στις Βρυξέλλες ήταν αποτέλεσμα θεσμικής απόφασης. Θέλαμε να επιτρέψουμε τη μεταφορά συνηθισμένων εργασιών, επικοινωνίας, ενημέρωσης κλπ. Ενημέρωσης πελατών, χρηστών οργανώσεων σε ευρύ τομεί από εκεί. Τρία χρόνια υπάρχει. Με διευθυντή, εποπτεία τριών γενικών διευθύνσεων, κυρίω για την κοινωνία των πληροφοριών, εκπαίδευση, παιδεία και έτκο, έδειξε ότι λειτουργεί σωστά. Τρία χρόνια είναι μια μέτρια περίοδος χρονικά, αλλά σε τρία χρόνια βλέπουμε πολλά αποτελέσματα στην πράξη όσον αφορά την ένταση της επικοινωνίας. Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισκέφθηκαν την υπηρεσία αυτή στα πλαίσια της θεσμικής συνεργασίας, κοντολογής. Πάνω από 22% του προπολογισμού ΑΕΑΚ για τον πολιτισμό και για την παιδεία περνάει από αυτό το φορέα. Ο διευθυντής, ο Ζίλμπετ είναι εδώ μαζί μας. Συγκρίνοντας αυτό με το κόστος των ιδίων προσπαθειών που καταβάλλονται από την ίδια τη Γενική Διεύθυνση, βλέπουμε ότι η απόδοση είναι 25% καλύτερη. Άρα σημαντικές οικονομίες και, και καλύτερη δουλειά βγαίνει. και οι γενικέ διευθύνσει ασχολούνται περισσότερο με την ε, πολιτική, διαμόρφωση πολιτική, προτεραιότητε πολιτικών, κεντρικέ δράσει, σημαντικέ εκδηλώσει, σημαντικέ δράσει. Και αυτό ευθυγραμμίζεται με την φιλοσοφία που ενστερνίζεται και το Κοινοβούλιο όσον αφορά το τι πρέπει να κάνουν αυτές οι υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζήπε. Ορίστε. Ναι, να πω κάτι άλλο πέρα από τα οικονομικά ωφέλη που έθιξε ο Επίτροπος. Νομίζω ότι οι δράσεις της υπηρεσίας στρέφονται γύρω από τρεις τομείς, κυρίως την ενίσχυση της διαφάνειας, αύξηση της διαφανείας και οι ιδιωτικοί φορείς να υπομισθούν περισσότερες ευθύνες και βέβαια και ενίσχυση των εσωτερικών ελέγχων και η σωστή διαχείριση των οικονομικών. Δεύτερη πτυχή, όλε οι δράσει απλούστευση όσον αφορά τα προγράμματα που αφορούν του πολίτε, με επιδοτήσει που πολύ συχνά είναι επιδοτήσει χαμηλέ, με χρήση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρει αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού δημιουργία εταιρικών σχέσεων ε, κατά καταβολή ε, ποσών που ενθαρρύνει το ελεκτικό συνέδριο και άλλοι παρόμοιοι μηχανισμοί που αφορούν την απλούστευση εφαρμόζονται. Τρίτον, Θέλουμε να δώσουμε τις καλύτερες υπηρεσίες στους δικαιούχους των επιδοτήσεων. Η έρευνα που έγινε πάνω σε 2.000 δικαιούχους για την αξιολόγηση της πρώτης τριετίας λειτουργίας της υπηρεσίας καταδεικνύει ότι μέσω δημόσιου φορέα και όχι ιδιωτικού φορέα όπως είναι το, ήταν η υπηρεσία ε, παροχής βοηθείας κατά το παρελθόν δείχνει ότι έχουμε βελτίωση όσον αφορά την εκτέλεση των δράσεων και όσον αφορά και την παρακολούθηση του τι γίνεται όσον αφορά τα χρήματα που χορηγούνται προς όφελος των δικαιούχων. Ευχαριστώ λέει ο κ. Σοντή για αυτές τις απαντήσεις οι οποίες είναι σαφέστατες. Πριν σας παρακαλέσω να ολοκλώσουμε τη Γενική Πτυχή κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σκέφτεστε για τις προκαταρκτικές δηλώσεις που εγκρίνατε όσον αφορά τις 39 εκτορικούς ε, οργανισμούς. Έχετε ένα από 329, μια επιφύλαξη πάνω 329, αλλά το συνέδριο είπε ότι δεν έχετε εισαγάγει τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης που θα έπρεπε να είχατε εισαγάγει βάσει της συμβατικές σχέσεις που έχετε με τις υπηρεσίες αυτές. Γιατί. Uh, Αυτό το σημείο καθορισμού αυτών των όρων, αυτών των κατηγοριών και που αφορούν ε, σημαντικές ε, συστάσεις ε, και που όσον αφορά τους αριθμούς σωρευτικά συνολικός αριθμός σε κάποιες περιπτώσεις είναι τρεις, άλλες είναι δεκατρεις έχουμε διαφορετικές καταστάσεις σε διαφορετικές υπηρεσίες, σε διαφορετικούς οργανισμούς. Όμως, κατά τα τέλη του 2008, Καμία από αυτές τις υποθέσεις δεν είχε χαρακτήρα τροχοπέδης ε, ή δεν ήταν τόσο σοβαρή υπόθεση ώστε να έπρεπε να σταματήσουμε τη χρηματοδότηση ή υποστήριξη αυτής ε, αυτών των οργανισμών. Εργαζόμαστε για αυτό τα πάνω σε αυτά τα ζητήματα για να βελτιώσουμε την κατάσταση για τους οργανισμούς και υπηρεσίες. Είχαμε συναντήσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Είχαμε 30 τρεις άμεσες επιτόπου επισκέψεις επιτήρησης ή εποπτείας σε αυτούς τους οργανισμούς. Έχουμε λοιπόν το ίμιση που επισκεφθήκαμε, στις υπόλοιπες θα τις επισκεφθούμε το 2009. Έλεγχοι οικονομικοί διοργανώνονται και η κατάσταση είναι συνολικά πολύ καλύτερη από ό,τι στο παρελθόν. Όταν ήρθα, σε αυτό τον τομέα, ζητήσατε να ακούσετε ποιες ήταν οι επιφυλάξεις. Έχουμε διάφορες αποφάσεις για την πάυση καταβολής κονδυλίων ή λειτουργία σε κάποια κράτη-μέλη. Έπρεπε να μεταμορφώσουμε το σύστημα από το παλαιό στο νέο. Δεν ήταν εύκολο πάντα να επεξηγούμε και να υπάρχει πάντα συμφωνία. Τώρα τις έχουμε και είναι γραπτές μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αποκεντρωμένων αυτών υπηρεσιών οργανισμών. Και για να καταφέρουμε τους εταίρους μας, τα Υπουργεία, στα κράτη-μέλη να επιμεριστούν την ευθύνη που τώρα έχουμε επιτύχει, είναι το αποτέλεσμα καθημερινής χειροπιαστής έμπρακτης δουλειάς με όλους τους οργανισμούς και υπηρεσίες, με όλα τα Υπουργεία και υπηρεσίες δεν είχαμε κάποια ε, σύμβαση ή συμφωνία που να έχουμε υπογράψει με οποιοδήποτε οργανισμό ή υπηρεσία προτού βεβαιωθούμε ότι τα μέτρα τα οποία είχαν υιοθετηθεί εφαρμοζόντουσαν με κάθε σοβαρότητα και ότι δεν θα υπήρχαν νομίζω προβλήματα αξιοπιστίας ε, ή επαγγελματικού χαρακτήρα για την ε, δυνατότητα υπογραφής τέτοιων συμφωνιών. Δεν είναι λοιπόν ένα τετέλεσμένο γεγονός μέρος μιας διαρκούς ενεξελίξη διαδικασίας αξιολόγησης και με ένα feedback αμφίδρομα αξιολόγησης. Τώρα το σύστημα λειτουργεί με βάση αμοιβέ συμφωνίες που βρίσκονται στη βάση τους και υπάρχει μεγάλη μίζων αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα 7 χρόνια ή τα προηγούμενα προγράμματα και τους ε, δημοσιονομικούς κανονισμούς. Ευχαριστώ. Τελειώνοντας, μπορείτε να μας πείτε τι σκέφτεστε γενικά μια που έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία και πρέπει μέχρι την να υποβάλουμε το κείμενο προς μετάφραση. Κατάλαβα ότι έχετε την εντύπωση ότι το σύστημα εξελίσσεται, αλλά εμείς βλέπουμε να υπάρχουν ποσοστά ασφάλματος της τάξης του 20%. Είναι τεράστιο αυτό. Τι σκέφτεστε για την ποιότητα διαχείρισης για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε μια καλύτερη εξολόγηση τη απαλλαγή. Uh, uh, Θα έλεγα γι' αυτό ολοκληρώνοντας το τέλος της εισαγωγικής μου παρατήρησης ότι βρισκόταν ευθυγραμμισμένο με τη γραμμή της, ε, του Ελληνικού Συνεδρίου διότι θεωρούμε ότι οι συστάσεις ή η μέρος ή το σύνολο που έχουν υλοποιηθεί στοχεύουν σε σημαντικούς στόχους και ποιοι είναι αυτοί είναι ο έλεγχος και το υποπτικό σύστημα που θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικά με την εφαρμογή αυτών των ε, εποπτικών ε, ελέγχων. Έχουν αναλυφθεί δράσεις λοιπόν και αυτά που βρίσκονται καθοδόν και όσον αφορά το 2008 και ιδιαίτερα τώρα στην, στην αρχή του 2009 και εφ' θα μπορούν να οδηγήσουν στο να εφαρμοστεί αυτή η προσέγγιση του συστήματος με αυτόν τον τρόπο. Να βασιζόμαστε με τις δηλώσεις αυτές και να έχουμε αξιόπιστη υλοποίηση και εφαρμογή υπό δημοσιονομικό πρίσμα ή διοικητικό πρίσμα στον τομέα του πολιτισμού και της παιδείας και εκπαίδευσης, κατάρτισης. Γνωρίζω ότι αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο υπό πολιτικό πρίσμα, αλλά και χρηματοοικονομικά. Κάνουμε λόγο για παραπάνω από ένα δις ευρώ ετήσια σχετικά με τον τομέα αυτό. Και θέλουμε σίγουρα να ευθυγραμμιστούν όλες αυτές οι αρχές με τις ε, αρχές ε, της, ε, του δημοσιονομικού κανονισμού και των νομικών βάσεων. Και συγκρίνοντας τους αριθμούς από τους υπολογισμούς και από την έκθεση το ε, έχει 15% έχουμε και αύξηση σε 45% των, ε, της επικοινωνίας όσον αφορά την Γενική Διεύθυνση. Η συνεισφορά της Γενικής Διεύθυνσης ΕΑΚ στο κεφάλαιο 9 το, της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι πολύ σημαντική υπό το πρίσμα της θετικής απήχησης ή την ε, ε, θετική αυτή πτυχή. Εργαζόμαστε στο τελευταίο τμήμα αυτής της ε, ενότητας και είναι θέμα δικής μου αρμοδιότητας και για την εξάντα δυνατότητα σύνταξης ε, ε, διασφαλίσεων από τα κράτη-μέλη το σύστημα λειτουργεί, οι κατευθυντήρες γραμμές έχουν υιοθετηθεί, οι εταίροι συνεργάζονται πλήρως και τούτων λεχθέντων νομίζω ότι μπορούμε να αναμείνουμε βελτιώσεις που θα σημειωθούν κατά τη διάρκεια του 2009 και του, της χωρίς απαλλαγής για το 2008. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Δεν έχω άλλες ερωτήσεις πρόεδρε. Σε ευχαριστούμε. Ο κύριος Λιμπεράτσκι παρακαλώ. Σας ευχαριστώ θα ήθελα να προσθέσω την ερώτησή μου στην ερώτηση του κυρίου Οντή πιο πριν. Επρόκειτο για 20% σφάρμα, ποσοστό σφάρματος και για 6.000 τέτοιους ελέγχους ε, ή τέτοιες δράσεις η αξιολόγηση τέτοιου ποσοστού σφάλματος είναι αξιόπιστη. Κύριε Επίτροπε, καταδείξτε μας, αποδείξτε πώς ε, υιοθετούνται και καταλήγουμε σε αυτές τις δειγματοληπτικές ε, δράσεις. Μπορούν να υπάρχουν διαφορετικές τέτοιες ε, δειγματοληπτικές δράσεις σε διαφορετικούς τομείς, σε διαφορετικά κράτη. Έχουμε 27 κράτη-μέλη, 150 τέτοιες δειγματοληπτικοί έλεγχοι και μοιράζονται ανακράτως πώς καθορίζονται αυτές οι δειγματοληπτικές δράσεις. Και δεύτερη ερώτηση κύριε Επίτροπε, ποια είναι η άποψή σας για την αποτελεσματικότητα των δαπανών. Κάθε ευρώ που δαπανάτε φέρνει κάποια πρόσθετη αξία δαπανάτε με αποτελεσματικό τρόπο, υπάρχει όφελος από αυτή τη δαπάνη. Αυτή η τάση είναι σταθερή και μόνιμη όσον αφορά την δημιουργία ωφέλους και όσον αφορά το συσχετισμό δαπανών και ωφελημάτων. Με άλλα λόγια, πώς διασφαλίζεται και ποια είναι τα ωφέλη των δαπανών σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι το πρώτο ερώτημα αφορά περισσότερο το ελεγκτικό συνέδριο και όχι εμένα όσον αφορά το ποσοστό ή τον τρόπο μετρήσεως του ποσοστιαίου σφάλματος και πώς αποφασίζεται αυτό και πώς μπορεί να βελτιωθεί. Σημαντικότερο νομίζω είναι το πώς να χρησιμοποιούμε τους πόρους για να πετευθούν οι στόχοι του προγράμματος με αποτελεσματικότητα, με διαφάνεια και νομίζω ότι αυτό είναι κοινό καθήκον. Αυτό που άλλαξε, όπως τα βλέπουμε εμείς τα πράγματα, σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως συγκεκριμένη Γενική Διεύθυνση, είναι το διοικητικό κόστος για την εκτέλεση των προγραμμάτων. Μειώθηκε από 8,9% σε 8,5% ε, σχεδόν ε, μία ποσοστία μονάδα λόγω εσωτερικής μεταρρύθμισης εν μέρη στη Γενική Διεύθυνση μετά λόγω της εισαγωγής της εκτελεστικής υπηρεσίας στο όλο σύστημα και λόγω των προγραμμάτων που αποφασίζονται. Είναι μια συνεχής πρόκληση αυτή να χρησιμοποιούμε τα χρήματα αποτελεσματικά. Κυρίως στους τομείς αυτούς όπου ασχολούμαστε με μεμονωμένους πολίτες και με την κινητικότητά τους. Και θέλουμε να δημιουργηθεί ένα συνέστημα συμμετοχής, πρόσβασης στα ευρωπαϊκά προγράμματα και πολιτικές και αυτό ανταποδίδει. Υπάρχουν πολλές θετικές αντιδράσεις όσον αφορά το μέλλον της Ευρώπης και τη συμμετοχή στο ευρωπαϊκό γίγναστο. Θα ήθελα να υπογραμμίσω λοιπόν τη μείωση των λειτουργικών εξόδων μείωση των προσθέτων δαπανών για τους χρήστες παραδείγματος χάρη πριν χρειαζόμασταν περιπλοκότερες διαδικασίες για τις αιτήσει. Τώρα που στέθηκαν τα πράγματα. Συντομότερες αιτήσει. Χρησιμοποιούνται περισσότερο τα καταποκοπήν ποσά πιο πολύ τώρα από ό,τι κατά παρελθόν. Και ο περίπλοκος τρόπος αξιολογήσεως επιλεξιμότητας εφαρμοζόταν παλιά. Τώρα αντί συμφωνιών για απλά προγράμματα παίρνουμε αποφάσεις για ε, υποτροφίες, για την χορηγία ποσών. Δεν χρειάζεται υπογραφή και των δύο πλευρών, αλλά απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολλά γίνονται άμεσα, μέσω υπολογιστού, online. Δεν χρειάζεται να στείλει την αίτηση ο ετών και να περιμένει. Χρησιμοποιεί τον υπολογιστή και ξέρει πολύ γρήγορα αν είναι επιλέξιμος ή όχι. Λαμβάνονται λοιπόν δέους αποφάσεις. Έχει λόγω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της προθυμίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της θετικής προσέγγισης, έχουμε μειώσει τον περίπλοκο χαρακτήρα της επιτροπολογίας. Και αυτό δείχνει αποτελεσματικότητα. Εξοικονομούμε χρόνο, χρήματα. Δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες για τους χρήστες. Για να μπορούν να χρησιμοποιούν τα χρήματα. Αυτή είναι η απάντησή μου. Και όσον αφορά την αξιολόγηση, αυτό είναι κάτι που αφορά περισσότερο το ελεκτικό συνέδριο. Λέβινσον έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ και ο καθηγητής Μπονίτσι είπαμε ότι πραγματικά πιστεύουμε ότι ε, τα είπαμε όλα σε αυτή την έκθεση. Δώσαμε πολλές πληροφορίες όσον αφορά τα πορίσματά μας. Τα σφάλματα που βρήκαμε στις διάφορους τομείς. Πίνακα 9.1 και πίνακα 9.2. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες. Περισσότερες από αυτές που δώσαμε κατά το παρελθόν. Δύο πράγματα λοιπόν. Δίνουμε πολλές πληροφορίες σε αυτό το κεφάλαιο. Και τελικά διαπιστώνουμε ότι οι δοκιμές που γίνανε και η δηματοληψία ανταποκρίνονται στις διεθνείς προδιαγραφές. Ο κύριος Χάρης έχει το λόγο. you, Σε ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Επίτροπο Φίγερ και σε σχέση με την συνεργασία για αυτά τα θέματα τα τελευταία πέντε χρόνια νομίζω ότι είναι εξαιρετική και είναι η ε, στοχοθέτηση να υπάρξει αποτέλεσμα για την χρήση των κονδυλίων των φορολογουμένων. Πρώτα απ' όλα όμως θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχω πρόβλημα να ησυχάσω και να κοιμηθώ το βράδυ και διαβάζω έτσι τις εκθέσεις του ε, ελεγκτικού συνεδρίου σε αυτό το εκτεταμένο κεφάλαιο 9 δεν μπόρεσα να βρω τίποτα που να δείχνει αν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι που γίνονται γίνονται με βάση οποιαδήποτε κατά προσέγγιση ad hoc ε, σε σχέση με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Υπάρχουν εδώ και ε, μεγαλύτερα δείγματα αλλά μικρότερα που ε, δημιουργούν και ζητήματα όσον αφορά τις ε, δειγματοληπτικές αυτές δράσεις του ε, συνεδρίου. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω το εξής. Μια και εξετάζοντας ξανά πράγματα όπως παλαιότερες εκθέσεις του ελεκτικού συνεδρίου ένα πράγμα το οποίο από πλευρά ε, της, ε, του Επιτρόπου ε, θα ήθελα να εξεταστεί σε σχέση με τις, τους ελέγχους εξ είναι κατά πόσον βλέπουμε ότι δίνεται μεγαλύτερη σημασία σε αυτές τις δράσεις εξάντε και ενώ γνωρίζω ότι είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να εξετάζεται είναι, έχει τη σημασία του. Ίσως θα έπρεπε να έχει τη συγκεκριμένη αυτή σημασία του σε σχέση με τις δράσεις του συνεδρίου. Κάποιες παρατηρήσεις, κάποια σχόλια για την διαβίου εκπαίδευση ε, το σχετικό πρόγραμμα. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που μου στείλατε τα παρατήματα και ερωτήματα για τα διάφορα ποσά που δόθηκαν στις διάφορες οργανώσεις και τα λοιπά τα εκτιμώ ιδιαίτερα αυτά από πλευρά σας. Εξετάζοντας κάποια ποσά και τους, τα αριθμητικά μεγέθη παρατηρώ ότι ένας αριθμός από αυτά τα προγράμματα θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν ούτως ή άλλως από εθνικές αρχές ή υπηρεσίες. Υπάρχει τρόπος να ελεγχθεί ότι δεν υποκαθιστούν τα δικά σας κονδύλια, κονδύλια τα οποία θα δινόντουσαν ή θα έπρεπε να δίνονται από εθνικές υπηρεσίες ή από πλευράς Υπουργείων στα κράτη-μέλη. Δεύτερον, υπάρχουν πολλές οργανώσεις που ε, σε σχέση με τους ελέγχους ε, στα κράτη-μέλη και που όσον αφορά τη διδημοποίηση πόλεων ή τα πανεπιστήμια. Τι γίνεται για πανευρωπαϊκές όμως οργανώσεις. Ποιο κράτος μέλος ε, είναι εκείνο το οποίο ε, έχει κάποια συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Το κράτος της έδρας ε, τέτοιων οργανώσεων ή και γνωρίζοντας ότι για παράδειγμα υπάρχουν κάποιες ενώσεις και σύλλογοι που έχουν ε, την έδρα τους σε ένα κράτος και δρούν σε άλλα και πέρα από ε, το κράτος έδρας τους. Κάτι σχετικό. Τι γίνεται λοιπόν εδώ. Και υπό το φως της ε, ευρωπαϊκής oh της ευρωπαϊκής αδελφοποίησης υπό την αντίστοιχη κατηγορία του προπολογισμού. Είναι, θα έλεγα, η κατηγοριοποίηση των ε, διδήμων αδελφών πόλεων. Πώς ε, όλα αυτά τροφοδοτούνται σε εσά για την εξέλιξη αυτών των πρωτοβουλειών και εκδηλώσεων ε, για να αξιολογούνται αν αξίζουν τον κόπο ή όχι. Πώς αξιολογείται η ποιότητα και ποιος έλεγχος υπάρχει για την, το αξιόλογο τέτοιων δράσεων. Και τελικά και ένα γενικότερο σχόλιο που ως ε, ευρωσκεπτικιστής θα αναμενόταν από πλευράς μου ίσως. Ε, εδώ σε σχέση με τα ποσά, τα κονδύλια τα οποία ε, καταβάλλονται. Λέει εδώ ανακοίνωση για την ευρωπαϊκή ενοποίηση και διάφορα άλλα σχετικά. Θα έλεγα είναι τα κονδύλια ή ε, τα θέματα για την ε, διαφήμιση, η προπαγάνδα αυτών των ε, δράσεων. Και εδώ υπάρχουν συναφή προβλήματα. Κάποια, κάποιες οργανώσεις είναι πολύ ικανές για να δρουν στο επίπεδο της διαβίου εκπαίδευσης αλλά εδώ θα έπρεπε να είμαστε πιο προσεκτικοί σε σχέση με τα διαφορετικά κριτήρια τα οποία θα απαιτούνται για να δίνονται τέτοια κονδύλια σε σχέση με ε, οργανώσεις ιδρύματα, να υπάρχει μια θετική συνιστόσα, ας το πω έτσι, ευρωπαϊκών δράσεων. Διερωτώ με λοιπόν σχετικά πόσα αυτά τα πράγματα έχουν τώρα και σε σχέση με τον προϋπολογισμό για να δίνονται κονδύλια θα πρέπει να υπάρχει η ε, επίδειξη, τέλο η αναφορά της, ε, του ευρωπαϊκού χαρακτήρα μιας τέτοιας δράσης. Αυτό ισχύει για όλα αυτά τα κονδύλια. Τι συμβαίνει. Για το πρώτο ερώτημα... <clears throat> Καλό θα ήταν το ελεγκτικό συνέδριο να τοποθετηθεί πρώτα, μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Μπονίτσι, παρακαλώ. Yes, thank you, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην παράγραφο 9.5α, στο κεφάλαιο τι βλέπουμε ότι βασιζόμαστε στην ουσιαστική ε, δοκιμή αντιπροσωπευτικού στατιστικού δείγματος 150 πληρωμών. Δεν είναι ad hoc. Βασίζεται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα. Βάση δειγματοληψίας μονάδων. Λαμβάνουμε υπόψη λοιπόν το μέγεθος. Μεγαλύτερες πληρωμές έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιλεγούν σε πρώτερες συζητήσεις κάποια μέλη αναφέρθηκαν στο σφάλμα του 21%. Αυτό είναι σφαλμένο. Είναι η συχνότητα των σφαλμάτων που είναι 21%, όχι το επίπεδο των σφαλμάτων. Τρίτον, το μέγεθος του πληθυσμού δεν σχετίζεται τόσο πολύ με το μέγεθος του δείγματος. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Μη συγχαίουμε τα δύο στοιχεία. 150 δεν είναι μικρό δείγμα. Μικρό δείγμα θα ήταν 30 ή λιγότερο. Τώρα αν είναι αρκετά αντιπροσωπευτικό το λαμβάνουμε υπόψη βλέποντας το επίπεδο εμπιστοσύνη. Εν τη αυτή περιπτώση έχουμε επαρκή εμπιστοσύνη και πιστεύουμε ότι το ποσοστό του σφάλματος είναι μεταξύ 2 και 5%. Και γιατί δίνουμε ένα φάσμα. Διότι είμαστε, έχουμε εμπιστοσύνη για το φάσμα αλλά όχι συγκεκριμένη τιμή, συγκεκριμένο ποσοστό. Αν θέλατε συγκεκριμένο ποσοστό θα χρειαζόσαστε μεγαλύτερο δείγμα για τους δικούς μας σκοπούς δοθέντες του μεγέθους του τομέα θεωρείται αξιόπιστο αυτό το φάσμα. Τέλος πριν από δύο χρόνια περίπου, είδα εδώ να κάνω, ήρθα να κάνω μια παρουσίαση για τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία. Ώρες πέρασαν. Συνέλεξα πληροφορίες και μπορώ να το κάνω ξανά αυτό αν κανείς όμως επαναξετάζει τα όσα εξετάστηκαν, δυσκολεύει η κατάσταση. Η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία πιστεύουμε ότι μας παρέχει αντιπροσωπευτικό αποτέλεσμα. Και είμαστε αρκετά διαθέσιμοι, μπορούμε έτσι σε ατομικό επίπεδο στην Επιτροπή εδώ να σας δείξουμε τι κάνουμε. Προφανώς μπορεί πάντα κανείς να βελτιώνει το επίπεδο της εμπιστοσύνης αλλά αυτό έχει κόστος. Ποιο είναι το κόστος. Χρειάζεσαι περισσότερους πόρους για να αναλύσεις τα στοιχεία, κάτι που μπορεί να κάνει δεχομένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι δεν χειριζόμαστε εμείς τα ποσά, εμείς ελέγχουμε τα ποσά αυτά. Οι διαχειριστές θα πρέπει να έχουν επαρκείς πληροφορίες και όπου υπάρχει πρόβλημα να έχουν επαρκή στοιχεία για να προβούν στη δέουσα διόρθωση και αν χρειάζεται να γίνει ανάκτηση ποσών. Άρα χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο εμπιστοσύνης και όχι μικρότερο. Ε, είναι ανοιχτή πρόσκληση αυτή, κύριε Πρόεδρε, να διεξαχθεί συζήτηση επί της μεθοδολογίας, διότι πιστεύω ότι στο κάτω-κάτω της γραφής πάντα επιστρέφουμε επί θεμάτων και αν το κάνουμε αυτό δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει την πρόοδο να πηγαίνουμε προς τα πίσω. Ο κύριος Φίγκελ. Ευχαριστώ Πρόεδρε θα ήθελα να πω ότι προετοιμάζοντας τα νέα προγράμματα διότι χρειάζεται διαπραγμάτευση για να επιτευχθεί συνένεση, να βρεθούν τα χρήματα με τις δημοσιονομικές αρχές. Πάντα φροντίζουμε να μην χρηματοδοτούμε αυτό που είναι ευθύνη των εθνικών ε, αρχών, αλλά να υποστηρίζουμε την ευρωπαϊκή δράση. Στα πλαίσια συνεργασίας, η χρηματοδότηση, Φερρυπίν, το Εράσμους αναφέρεται συχνά, να πω ότι πριν από μερικέ εβδομάδες τα κράτη-μέλη επενδύαν περισσότερα στην κινητικότητα ενώ εμεί επενδύαμε από, τον Ευρωπα... από ό,τι επενδύαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, προπολογισμό, σε εθνικό επίπεδο μέσω πανεπιστημίων γινόταν οι επενδύσεις. Δεν κινητοποιούμε πάντα άλλου πόρου. Υπάρχουν πάντα κάποια ανώτατα όρια όσον αφορά τη συγχρηματοδότηση. Αυτό δεν σημαίνει αντικατάσταση ευθυνών ή το να πληρώνουμε αυτό που είναι ευθύνη άλλων εθνικών ή τοπικών αρχών. Όσον αφορά τον έλεγχο, ε, το σύστημα αυτό έχει αποδειχτεί, εξαρτάται από τον ε, εταίρο, ακόμα και στην περίπτωση ευρωπαϊκών δικτύων ή πανευρωπαϊκών δικτύων και πανευρωπαϊκών φορέων, έχουν κάπου μία έδρα. Ένας εθνικός φορέας είναι ο στενότερος συμβατικός συνεργάτης. Αυτός ο φορέας λοιπόν ανάλογα με την έδρα του, το νομικό πλαίσιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον Επίτροπο ή την εκτελεστική υπηρεσία κινούνται. Ε, εμείς δραστηριοποιούμε θα υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν περιμένουμε. Είμαστε ενεργοί, πηγαίνουμε ad hoc, συνεργαζόμαστε με φορείς, αυτοί έχουν το δικό του σύστημα ελέγχου, ε, υποβάλλονται και εκθέσεις, όχι μόνο για την προετοιμασία μιας δράσης, αλλά και ενδιάμεσες εκθέσεις και τελικές εκθέσεις. Θα έλεγα ότι βασικά αυτό είναι ευθύνη των εθνικών αρχών, των εθνικών υπηρεσιών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των εκτελεστικών φορέων. Τέλος, το άκουσε δε στο ζήτημα της προπαγάνδας όπως των φορέων προπαγάνδας. Εγώ δεν θα χρησιμοποιούσα αυτή την ονομασία, τέλο πάντων. Αναφέρονται στη νομική βάση. Το πρόγραμμα για την ηθαγένεια, την ευρωπαϊκή υπηκότητα συμπεριλαμβάνει εννέα οργανισμούς που αναφέρονται συγκεκριμένα ως εταίροι. Υπάρχει ο κατάλογος. Είναι ευρωπαϊκοί φορείς που αναμειγνύονται στον τομέα της ενημέρωσης, της έρευνας, παιδείας, της εκπαίδευσης, μελέτης ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως το Ίδρυμα, η Ένωση ε, Jean Monnet, το Centre Européen Schumann και παρόμοιοι φορεί που έχουν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο, αυτό το Κοινοβούλιο. Και άλλα κινήματα, το ευρωπαϊκό κίνημα. Τι προτείναμε λοιπόν, ένα κομμάτι της τωρινής λύσης, σταδιακή εκπνοή, να μην υπάρχει προσήμιωση για το μέλλον. Η απάντησή μου ποια είναι ότι αυτή η πρακτική λίγη το 2009 και το 2010 και πέρα όλοι οι φορείς θα πρέπει να ανταγωνίζονται όπως όλοι οι άλλοι για να τύχουν υποστηρίξους. Αυτή είναι νέα προσέγγιση. Πιο ανοιχτή. Περισσότερες δυνατότητες για νέους φορείς. Χρειαζόμαστε όμως και καλά δίκτυα, παλιά δίκτυα όπου ξέρουμε περί τίνος πρόκειται και τι θα γίνει σε 10, 20 ή 50 χρόνια. Και θα είναι πιο ανοιχτέ ευκαιρίε για όλου. Να υπογραμμίσω αυτό που είπατε στην αρχή για τη συνεργασία τη δική μα. Πέρσι υπογράψαμε χορηγία για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Πικότητα και την Ευρωπαϊκή Παραλυμπιακή Επιτροπή για να υποστηρίξουμε τα άτομα με αναπηρία στον αθλητισμό. Είναι καλό για ένταξη, για συμμετοχή, αυτό ε, για πολλά, για πολλέ αξίε που πρέπει να υποστηριχθούν και στην Ευρώπη και στον κόσμο για τον αθλητισμό και για την ευθύνη. Οι ειδικέ, οι ειδικοί Ολυμπιακοί αγώνε λοιπόν, που ζητούν υποστήριξη. Και αν προβλεφθεί ειδικό κονδύλιο από το Κοινοβούλιο, θα ασχοληθούμε με αυτού του φορεί. Ο ρόλο μα είναι να δημιουργούμε δυνατότητε. Δικαιοσύνη, ανοιχτή προσέγγιση. Και πώ το πετυχαίνουμε αυτό. Αυτό είναι δική μας ευθύνη πώς το επιτυχίνουμε. Λοιπόν, κάτι έχει εγκριθεί συγκεκριμένα άμεσα στο πρόγραμμα. Κάτι άλλο στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων, κάτι προβλέπεται στα ειδικά κονδύλια του Κοινοβουλίου όταν εγκρίνει τον ετήσιο προπολογισμό, αλλά η τάση τώρα είναι επικοδομητική, είναι θετική. Δικός μας ρόλος είναι να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τα πράγματα, να είμαστε πιο ανοιχτοί. Ήδη όμως έχει επιτευχθεί η αλλαγή και αν χρειάζεται χρειάζονται και άλλε πληροφορίε. Είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε πολλέ πληροφορίε στα παραρτήματα, πληροφορίε που ζητήσατε. Το ζητήσατε αυτό, έχετε το κείμενο, μπορούμε να μοιραστούμε μαζί σας και λεπτομέρειε για όλες τις δράσεις που έχουν εγκριθεί, αν το θέλετε. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκρέσλε παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό που είπε ο Επίτροπος πιο πριν και να ρωτήσω σχετικά ποιες επιπτώσεις έχει η αναθεωρημένη δημοσιονομική, ε, δημοσιονομικός, δημοσιονομικός κανονισμός στο χαρτοφυλάκιο. Κάτι είπε για απλουστεύσεις ε, και αποτελεσματικότητα. Θα ήθελα να ακούσω περισσότερες λεπτομέρειες. Ποια είναι η πείρα που έχει συλλέξει με τον αναθεωρημένο αυτό δημοσιονομικό κανονισμό στο έργο του. Η δεύτερη ερώτηση αφορά το, τις διοικητικές δαπάνες. Έχουμε ήδη πέρυσι ρωτήσει ποια είναι, ποιες είναι οι διοικητικές δαπάνες. Μειώθηκαν πράγματι αυτές οι διοικητικές δαπάνες. Τώρα με ενδιαφέρει αν ο Επίτροπος προβλέπει περαιτέρω μείωση που θα είναι εφικτή αυτών των ε, διοικητικών δαπανών. 13,2-13,8% σε αυτό το ύψος οι δικτύες δαπάνες είναι, στο οποίο βρίσκονται είναι πολύ ψηλέ. Θα με ενδιαφέρε να ακούσω ποια είναι η πρόοδος που μπορεί να προαναγγείλει ο Επίτροπος για το μέλλον για τη μείωση αυτών των δαπανών. Υπάρχει μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αποδεκτό λέει κίνδυνο σε σχέση με τέτοιου είδου δαπάνε. Ο πολιτισμό όμω δεν συμπεριλαμβάνεται ούτε και στην στη συνοπτική κατηγορία, στον πίνακα για το, τα κόστη. Με ενδιαφέρει να γνωρίζω γιατί συμβαίνει αυτό. Επίση, γιατί η διαβίου εκπαίδευση δεν βρίσκεται πια εξειδικευμένα σε αυτά τα στοιχεία σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη. Θα με ενδιαφέραν τα αριθμητικά μεγέθη της διαβίου εκπαίδευσης τους αριθμούς αν μπορούμε να τους έχουμε και για την χρηματοδότηση μη κυβερνητικών οργανώσεων για το παράρτημα στις γραπτές ερωτήσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω αν κάπου και αν ναι, σε ποιο πρόγραμμα και περίπου σε ποιο αριθμητικό μέγεθος, ποιος είναι ο αριθμός ε, των ε, δαπανών για τη χρηματοδότηση αυτών των ΜΚΟ. Ευχαριστώ. Um, Μάλιστα, Πρόεδρε. Δημοσιονομικός λοιπόν, κανονισμός, νομίζω, τώρα έχει οριμάσει, αν θέλετε, περισσότερο. Είναι πιο φιλικός προς το χρήστη, επιτρέπει στους οργανισμούς να είναι πιο κατάφυστος στους πολίτες, πιο ευέλικτος και να ανταποκρίνουν καλύτερα ανάγκες της Ευρώπης. χαιρετίζω την είναι αυτή η προσέγγιση. Γιατί όταν εγώ άρχισα να με το τομέα αυτό, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλέ δυσκολίε από το παρελθόν. Ο κ. Σιτών Χάρη ήδη αναφέρθηκε στο 1999 και την κατάσταση τότε. Το αισθάνθηκα πάρα πολύ έντονα και κάναμε πολλές προσαρμογές των οποίων τους καρπούς τρέπουμε ε, τώρα κάνει να υπάρχει περισσότερη εμπιστοσύνη, υποστήριξη για το φυλάκιο αυτό. Η εκπαίδευση είναι σημαντική, αλλά υπάρχει και μεγαλύτερη ε, εμπιστοσύνη. Ε, να μου ζητήσει να ασχοληθώ με το IT που πιστεύουμε ότι είναι ακριβωμένο αλλά χρήσιμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά για το μέλλον της Ευρώπης ακριβώς αυτή η εμπιστοσύνη που αναπτύσσεται, που, που αυξάνεται και που καλύπτει όλους τους τομείς και τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις. Όσον αφορά λοιπόν το δημοσιονομικό κανονισμό και τη νέα νομική βάση, μας επιτρέπει κατά βάση μία απλούστευση. Αυτό είναι η πιο ορατή καινοτομία. Τα έντυπα υποβολή ε, ενδιαφέροντος είναι πιο απλά, πιο σύντομα. Έχουμε και νέες δομές εφαρμογής όπως σας είπα προηγουμένως γιατί αναδιοργανώσαμε τις εθνικές υπηρεσίες και ε, εγκαθιδρύσαμε πολιτιστικά σημεία επαφής, ε, εισαγάγαμε μόνιμους οδηγούς προγράμματος, χρειάζεται λιγότερος χρόνος για να αξιολογηθεί η κατάσταση, μειώνονται πολλές βαριές διαδικασίες επιτροπολογίας, επιτέθηκε αυτό λόγω και συνένεση του Κοινοβουλίου, είναι κατά είναι ποσά, αυτή είναι μια πρακτική που θα πάει και ευρύτερα χρησιμοποιείται. Εγώ αναφέρθηκα στην αυξανόμενη χρήση των αποφάσεων της Κομισιόν και όχι συμφωνιών, πράγμα που στην μήνυ δικασία κατά μέχρι και δύο εβδομάδες. Τώρα συγγνώμη, υπογράφουμε πολυετή συμφωνίες για τη χορήγηση των ποσών αυτών. Όλα αυτά λέω επειδή μας τα επιτρέπει και ο, ο Δημοσιονομικός και η νομική του βάση. Η απλούστευση αυτή δηλαδή είναι έτσι σημαντική. Είπα προηγουμένως ότι η προσημείωση σιγά σιγά εξαλείφεται και αυτό είναι ένα σημείο της καταρχήν συμφωνίας ε, της αρχής της θητείας αυτής και είναι σε προς νομίζω όλων. Διοικητικό κόστος τώρα, κατά πόσο είναι δυνατόν να έχουμε κατά νου περαιτέρω μείωση, ναι. Καταρχήν, ναι. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι περαιτέρω και πιο ομαλή λειτουργία των προγραμμάτων που άρχισαν το 2007. Το πρώτο έτος είναι πάντα πιο δύσκολο, πιο ιδιάζωνο θέλετε. Από εκεί και πέρα έχουμε μια συνοχή που θα πρέπει να οδηγήσει σε πιο ομαλή λειτουργία. Επίσης προετοιμασία μελλοντικών αναθεωρήσεων του προγράμματος και μπορούμε εκεί να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στις αδελαμίες. Μπορούμε να αποκομίσουμε νομίζω διδάγματα από πιο επιτυχείς ε, τομείς όπως η εκπαίδευση, η διαμήρη εκμάθηση. Οι εμπειρίες που είχαμε εκεί μπορούν να μεταφερθούν σε άλλα προγράμματα. έχουμε τέσσερα προγράμματα για βιοεκμάθηση, ηθαγένεια, πολιτισμός και νεολαία. Θα υπάρχουν στο μέλλον περισσότερες ε, επιχορηγήσεις μεμονωμένα, ιδίως στον τομέα της νεολαίας. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ε, αρέσει η προσέγγιση του να αναπτύσσεται ένας αποδεκτός κίνδυνος. Και η θέση της Κομισιόν είναι αυτή από το του περισμένου έντος. Θα πρέπει να το συζητήσουμε μεταξύ Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Εκτελεστικής Επιτροπής και να συμφωνήσουμε στον ορισμό και στον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε και συμπεριλαμβάνουμε αυτόν τον αποδεκτό κίνδυνο στους τομείς που μας απασχολούν. Τα σχέδια κινητικότητας τώρα οπωσδήποτε έχουν λιγότερο διοικητικό κόστος από ότι άλλες μεγάλες και συγκεκριμένες δράσεις. που δεν είναι πανταληπτικές, αν θέλετε. Αυτό που πιστεύω είναι ότι έχουμε εδώ μία από τις σημαντικότερες ε, πολιτιστικές ε, ή γενικά δράσεις ε, το Νοέμβριο, ότι συμφώνησαν και οι 27 υπουργοί ότι θέλουμε η κινητικότητα των νέων να είναι ο κανόνας, όχι η εξαίρεση. Απέχουμε βέβαια. Η σημερινή πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική, αλλά αν υπάρχει αυτό το όραμα να πραγματοποιηθεί μετά από 10-20 χρόνια, στο πως είναι πραγματικότερα. Το 87 το Ορασμούς ε, είχε καταδικαστεί από πολλούς. Γιατί υποβάλλει τέτοιο πρόγραμμα η Κομισιόν ελέγχθη ε, χωρίς να υπάρχουν και τα χρήματα, αν υπάρχει τίποτα άλλο. Τώρα όλοι όμως είναι σύμφωνοι με το πρόγραμμα Ερασμός. Έχουμε και την διαδικασία της Πολώνια που κινητοποιήθηκε. Όλα αυτά βοήθησαν. Δεν λέω ότι ήταν θαυματουργό το πρόγραμμα Έρασμος, αλλά ήταν ένα μέσο που μας επέτρεψε τη σύνδεση, αν θέλετε, που μας επέτρεψε τα διάφορα συστήματά μας να γίνουν συμβατά και να επιτρέψουν μια πραγματική κινητικότητα των πολιτών με διάφορες ικανότητες. Για τις μη κυβερνικές οργανώσεις αυτό το κατάλογο αυτό που κάναμε είναι ότι όπως μας ζητήθηκε εξαιρέσαμε τις σχολές και τα πανεπιστήμια. Όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν στο κατάλογο αυτό. Αλλά δεν είναι όλες οι οργανώσεις αυτές τις μη κυβερνικές οργανώσεις. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο ορισμό του τι είναι η μη κυβερνική οργάνωση. Ίσως χρειάζεται για συγκεκριμένες ε, ε περιπτώσεις συγκεκριμένα θέματα, συγκεκριμένο κονδύλι, δαπάνης, αν θέλετε κάποια διευκρίνηση, μπορώ να επανέλθω γραπτά. Αλλά δεν έχουμε τίποτα το και καλυμμένο. Δεν υπάρχει καμία σάφια μέσα στα πλαίσια των προγραμμάτων. Η κυρία Γκρέσλα θέλει μια συμπληρωματική ερώτηση νομίζω. Ζήτησα να μου πείτε τι γίνεται για ε, την ενίσχυση της, του λειτουργικού κόστους ε, αυτών των ε, υπηρεσιών. Πού βρίσκεται αυτό σε αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή επιδοτούνται και υπάρχει η δυνατότητα στήριξης με τέτοιες επιδοτήσεις για το λειτουργικό τους κόστος. Ευχαριστώ. Το γνωρίζετε απ' έξω. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο να απαντήσετε. Στα προγράμματα αυτά δίνουμε δύο ειδών ενισχύσει. Από τη μία πλευρά ενισχύσει προγραμμάτων για συγκεκριμένο στόχο και για αυτά τα προγράμματα δίνουμε και επιδοτήσεις λειτουργίας αν θέλετε. Operating grants. Σπληρούνται κάποια κριτήρια ε, κατανομής και επιλεξιμότητας ενώσεις που έχουν συγκεκριμένο στόχο και ευρωπαϊκό σκοπό και δίνουμε μια κάλυψη που καθορίζεται τη βασική νομική βάση μέχρι ένα ποσοστό των διοικητικών δαπανών διαχείρισης αυτών των οργανισμών. Από τη στιγμή το πρόγραμμα εργασίας τους βεβαίως αντιστοιχεί στους σκοπούς του προγράμματος και στα κριτήρια κατανομή σύμφωνα με την ε, πρόταση. Πάντα όπως την υπογράμμισε και ο Ευρωπαϊκός Επίτροπος μάλλον μέσω διαδικασίας ε, προσκλήσεως υποβολής προτάσεων. Ενδιαφέρον θα ήταν ακριβώς για μας να γνωρίζουμε ποια είναι αυτά και να έχουμε και ένα ποσοστό του συνολικού δηλαδή κόστους για τις επιδοτήσεις αυτές. Είναι δυνατόν να γίνει αυτό ή είναι μεγάλη, ε, μεγάλο, πολύ, μεγάλη, πολύ μεγάλο διοικητικό πρόβλημα να μας το δώσετε. Όχι, όχι. Είναι δυνατόν να σας δώσω για τα συγκεκριμένα προγράμματα και για την παιδεία και τον πολιτισμό, νεολαία, ηθαγένεια, σας δώσουμε τα ποσοστά που αφορούν την επιδότηση του κόστους λειτουργίας. Μπορούμε γραπτώς να απαντήσουμε. Είναι αρκετά χαμηλό το ποσοστό για όλα τα προγράμματα εφόσον ο σκοπός πάνω απ' όλα είναι να ε, εγκριθούν, είναι ο σκοπός των προγραμμάτων και τα ονόματα των οργανισμών, λέει κύριε Κρέσλο. Μάλιστα. Ο κύριος έχει το λόγο. Uh, um, uh- Δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό. Να σας υπενθυμίσω διάφορες θεωρίες των κοινωνικών επιστημών. Ο κύριος Μπονίτσι, ο καθηγητής Μπονίτσι λέει ότι το τυχαίο δείγμα των 150 είναι μεγάλο, αρκετά μεγάλο, όχι μικρό. Μετά η θεωρία των, ε, αυτών που συμβαίνουν, των συνεπιών μάλλον. Να δούμε κατά πόσο τα χρήματα χρησιμοποιούνται για τον σκοπό. Ειλικρινός και αποτελεσματικός. Και κάτι άλλο. στο σχέδιο Μάρσελ, Δεκαετία, τέλος δεκαετία 40 και το 50. Ζήτησε η Αυστρία χρήματα για να φτιάξει την όπερα της Βιέννης. Και μας είπαν ότι το σχέδιο Μάρσαλ δεν είχε αυτό το σκοπό. Πήραν λοιπόν χρήματα από την κυβέρνηση για την επισκεφτή ιδεολεκτικών σταθμών στις Άλπεις και τα χρησιμοποίησαν τα χρήματα αυτά για την όπερα και ζήτησαν και για τον ιδιολεκτικό σταθμό χρήματα και τα πήραν σαν ενίσχυση του σχεδίου Μάρσαλ. Άρα, de facto, τα χρήματα του σχεδίου Μάρσαλ πήγαν για την όπερα. Δεν το ξέρουμε πότε θα γίνει έτσι. Το μόνο που είμαστε σίγουροι ότι αν τα χρήματα δίνουμε πάνω για έναν σκοπό για τον οποίο δεν θα τον ερευόταν να τα χρησιμοποιήσει αυτή η χώρα. Τότε αν γίνεται αυτό πάει 100% για το σκοπό. Μπορεί να πηγαίνουν τα χρήματα για κάτι που θα ήθελα να κάνω έτσι και αλλιώς και τα χρήματα μπορεί να πάνε για κάτι άλλο. Δεν είναι θέμα που αφορά τόσο πολύ την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού, αλλά όλο το Κοινοβούλιο που θα πρέπει να εξετάσει αυτό, αυτή τη θεωρία των συνεπειών και των αποτελεσμάτων. Όταν δίνουμε τα χρήματα για κάποιο σκοπό, πράγματι εκεί πάνε ή πάνε για κάτι εντελώ διαφορετικό. Και εγώ διατείνομαι ότι πηγαίνουν σε κάτι εντελώ διαφορετικό. Να παραμείνουμε όμως στο θέμα του κυρίου Φίγκερ στις παρεμβάσεις μας. Έχω γενικά κατανόηση για γενικά σχόλια. Κύριε Κάμερα, έχετε τον λόγο και μετά θα ολοκληρώσω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάνω στο τελευταίο που υπόθηκε. Κάτι που αφορά βασικά το ελεκτικό συνέδριο. Έχω ερώτηση. Υπάρχει κάποια εκτίμηση. Έλεγχος, όχι τόσο έλεγχος, αξιολόγηση. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της χρήσης αυτών των χρημάτων. Μπορεί να αποδειχτεί ότι οι αποδέκτες των χρημάτων δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, ότι βελτιώνουν την παραγωγικότητα μέσω των προγραμμάτων, η αποδοτικότητα κλπ. κλπ. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι αυτοί που παίρνουν τα χρήματα είναι χαρούμενοι. Το ερώτημά μου όμως, όπως και για άλλες δαπάνες Ευρωπαϊκής Ενώσεως, είναι τι παίρνουμε για τα χρήματά μας τελικά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα χρήματα αυτά βγαίνουν από τα κράτη-μέλη. Από ανθρώπους που θα τα χρησιμοποιήσαμε με διαφορετικό τρόπο. Τα παίρνουμε. και περισσότερε δαπάνε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω θα χρησιμοποιούνται διαφορετικά στα κράτη-μέλη. Τουλάχιστον στη χώρα μου δεν θα χρησιμοποιούσαμε χρήματα με αυτόν τον τρόπο που συζητάμε. Πώ κρίνουμε την αποτελεσματικότητα τη χρήση των πόρων που διαθέτουμε. Μου είπαν ότι θα πρέπει να, μια και έχουμε web streaming, να υπάρχει η δυνατότητα ε, αυτή της ε, παρέμβασης. Υπάρχουν απαντήσεις ε, από πλευρά του Επιτρόπου και από τον Γενικό Εισηγητή και μετά ολοκληρώνουμε. Κύριε Φίγκερ, θέλετε να παρέμβετε σύντομα, παρακαλώ. Yes, yes, Mr. President. Μάλιστα, Πρόεδρε, ίσως μπορείτε να προσθέσετε κάτι σε αυτιακό παράδειγμα. Λέω, μιλάει για τον Herbert Bosch που ήταν πρωταγωνιστής της διεύρυνσης. Γνωριζόμαστε χρόνια πριν την προσχώρηση της χώρας μου στην Ένωση. Η ευρωπαϊκή εμπειρία είναι σημαντικότατη για το μέλλον. Σχέδιο Μάρσαλ ή όχι, ένα σχόλιο. Η Τσεχοσλοβακία το 1947 εξέφρασε ενδιαφέρον να μπει, να ενταχθεί στο σχέδιο Μάρσαλ. 48, Φεβρουάριο του 48. Αντεστράφησαν τα πάντα. Και ο Στάλιν αποφάσισε ποιος μπαίνει και δεν μπαίνει. Ήμασταν στα χέρια του Στάλιν. Θα μας άρεσε να μπορούμε να παίξουμε αυτά τα χρήματα για την όπερα, για τα, να φέρουμε παρόμοια παραδείγματα για ηλεκτρικούς σταθμούς κλπ. Θα μπορούσαμε λοιπόν να είμαστε ιδρυτική χώρα διαφορετικά. Η ιστορία όμως δεν ασχολείται με υποθέσεις και θεωρίες. Λοιπόν, παιδεία, εκπαίδευση, δεν υπάρχουν επενδύσεις για υποδομές, αλλά είναι κινητικότητα, συνεργασία καλλιτεχνών. Δεν τα πάντα ρόδινα βέβαια. Ασχολούμαστε όμως με ανθρώπους, την εκπαίδευσή του, τα προσόντα τους, την αναγνώριση των γνώσεών τους, τη μεταφορά των γνώσεών τους, την ενσωμάτωση των γνώσεων στην πραγματική οικονομία επαφή ανθρώπων με ανθρώπους, ε, εορτασμούς που σκέφτονται και θυμίζουν τα θύματα του σταλινισμού και του ναζισμού. Κατά το παρελθόν, μετά το 1999, στο Κοινοβούλιο κυρίως, υιοθετήθηκαν κανόνες και προγράμματα όπου δεν προβλέπαμε εκεί ότι όλοι είναι απαταιώνες εμείς θεωρούμε ότι οι αποδέκτες είναι χρήστες τίμοι, ε, ειλικρινείς εταίροι. Εάν θεωρούμε κάτι διαφορετικό να το αποδείξουμε. Δεν ξεκινάμε την υπόνοια ότι όλοι είναι απαταιώνες. Κάτω παρελθόν ε, ε, αίτιο δυσκολιών ήταν αυτή η υπόθεση. Και υπήρξαν αρνητικές αντιδράσεις για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Δεν είναι όλα τέλεια τώρα. Ακολουθούμε όμως διαφορετική προσέγγιση. Και ήθελα να πω ότι εδώ μιλάμε για επιλεξιμότητα. Δηλαδή, συμμόρφωση με βασικά κριτήρια, έλεγχο, εποπτεία, αξιολόγηση. Και τέλος, εξίσου σημαντικό, ποια είναι η απάντηση όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη γενική αξιολόγηση ή την εξέλιξη των προγραμμάτων. Εκεί ετοιμάζουμε μια διάμεση αξιολόγηση και αναθεώρηση. Οπότε εδώ μπορούμε να εστιαστούμε περισσότερο στην κινητικότητα, πώς θα μειώσουμε τις δαπάνες, το διοικητικό κόστος και στο δεύτερο ερώτημα για τα αποτελέσματα, τα γενικά αποτελέσματα για μας, αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα ή σημεία, διότι αυτό που συμφωνούμε σε ευρύτερους τομείς πολιτικής, που είναι εθνικές πολιτικές, είναι κάτι που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα. Αν πιστεύουμε ότι η κινητικότητα είναι κάτι καλό, ότι η διεθνοποίηση των πανεπιστημίων μας η αναγνώριση πτυχίων και διπλωμάτων είναι σημαντικά, πρέπει να τα υποστηρίξουμε αυτά ως στόχους μέσω των καταλήλων εργαλείων. Και το πρόγραμμα είναι ένα εργαλείο για την υποστήριξη της συνεργασίας της διαδικασία της Μπολόνια Φερρυπίν. Και έχουμε δεύτερη διαδικασία αυτή της Κοπενχάγης για την επαγγελματική κατάρτιση. Πάντα ήταν στη σκιά των μεταρρυθμίσεων ή τη Μπολόνια. Χρειαζόμαστε όμω ανθρώπου με δεξιότητε. Και με την κρίση και χωρί την κρίση. Οι δεξιότητε σημαίνουν πολλά και τα προσόντα. Η διαβίω εκμάθηση κλπ. Και, και, και ούτω καθεξής. Δεν θέλω να πω τα πάντα είναι ξεκάθαρα, όμως η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και η γενική το γενικό αποτέλεσμα που επιτυχαίνει ένα πρόγραμμα για μας είναι πολύ σημαντικό και με τα χαρά συζητήσαμε με τον κύριο Λέβινσον. Και είδαμε ότι και το ελεκτικό συνέδριο παρόμοια προσέγγιση ακολουθεί. Βεβαίως δεν αμφισβητούμε τα βασικά στοιχεία, θα πρέπει η επιλεξιμότητα, η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα να παραμείνουν σαν όρια για την εκτέλεση του προγράμματος, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε επίσης και τι πετυχαίνουμε μέσω του προγράμματος. Και είναι πιο όρημη αυτή η προσέγγιση. Είναι πιο όρημη η κοινότητα. Μιλάμε για στόχους περισσότερο από ότι λεπτομέρειες. Είναι αλλαγή αν συγκρίνουμε την κατάσταση τωρινή με την κατάσταση πριν από αρκετά χρόνια. Και παλιές συζητήσεις εδώ, εγώ ήρθα το 2004 και... Αυτό εννοούμε, τις παλιέ συζητήσεις με τώρα. Ευχαριστώ. Πείτε. Κύριε Σιγητά, κάτι να προσθέσετε, παρακαλώ, Δεν έχω ερωτήσει, συγκεκριμένε ε, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τις απαντήσεις ε, που έδωσε, που είναι συγκεκριμένε και κρατά και προφορικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπο. Σας ευχαριστώ το ηλεκτρικό συνέδριο που είναι ένα βασικότατο σώμα των προβλημάτων που έχουμε εδώ. Χάρηκα που είχαμε την ανταλλαγή από στον αυτή για το δείγμα. Κατάλαβα ότι το 21% ήταν ο ρυθμός, όχι τα ποσά. Ε, Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τα διαρθρωτικά ταμεία, αναφερόμαστε 11% εκείνη τα ποσά, το 21% τώρα είναι ο αριθμός των σφαλμάτων. Ε, σημαντικά ποσά βέβαια, αλλά αυτά είναι θέματα που αρχίζουμε τώρα να εξετάζουμε με το πλαίσιο του ανοιχτού σφάλματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα κατά εξαίρεση, το ελεκτικό συνέδριο. Η τελευταία λέξη, κ. Λέβης. Uh, Ευχαριστώ. Ρωτήθηκε αν κάναμε κάποιους ελέγχους για την αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα κτλ. Μπορώ να απαντήσω ότι στο σύνολο είναι μια νέα παράγραφος ε, που έχουμε στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και έχουμε και μια νέα υπηρεσία στο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο που αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα. Ξεκινήσαμε τη δουλειά λοιπόν και έχουμε προχωρήσει. Δεν έχουμε όμως τελικά αποτελέσματα. Ελπίζω ότι θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια του 2009, ώστε θα επανέλθουμε για να απαντήσουμε αυτό. Θα ήθελα επίσης να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος ότι αυτό το νέο κεφάλαιο ουσιαστικά θα μπορούσε στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού να αποτελέσει να δώσει ε, την ευκαιρία συζήτησης αυτών των θεμάτων για δύο ώρες ε, απόδειξη ότι ενδιαφέρον, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα θέματα και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά. Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι φυσικά στον έλεγχο, στην έκθεσή μας λέμε ποια είναι τα αποτελέσματα και βρήκαμε ότι υπάρχει ποσό σφάλματος, υπάρχει ανάγκη βελτίωσης των ελέγχων και του εποπτικού συστήματος σίγουρα αλλά αυτό που προσπάθησα να πω είναι ότι έχω την εντύπωση ότι έχοντας δει τις απαντήσεις που δόθηκαν από τον Επίτροπο, από την Επιτροπή, ότι βρίσκονται στην ορθή κατεύθυνση. Αν υλοποιηθούν οι συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου, πράγμα που ελπίζω ότι θα γίνει και έτσι λοιπόν μετά τους ελέγχους μας θα επανέλθουμε του χρόνου για να σας πούμε το τι συνέβη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο τώρα. Και πάλι θα ήθελα να υπενθυμίσω κάτι και στην αρχή ίσως ήταν ίσως πολύ σύντομο ή δεν το ανέφερα ως πρόεδρος επαρκώς. Είναι αξιοπρόσεκτη ιστορία πρέπει να πω ότι με αυτό το ε, web streaming αυτή η πολιτική και η αξιολόγηση και ο έλεγχος αυτής της πολιτικής παγκόσμια ε, μπορεί να έχει απήχηση. Τώρα ποιος μπορεί να παρακολουθεί, ποιος παρακολουθεί όχι είναι άλλη υπόθεση. Δεν ε, είναι υποχρεωτικά ε, σε όλα τα κράτη-μέλη το ίδιο ενδιαφέρον. Είμαι όμως ευγνώμων για την δυνατότητα αυτή συζήτησης και παροχής αυτών των στοιχείων. Ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Γνωρίζω ότι έχουμε έναν συνάδελφο ο οποίος πιέζεται από πλευράς χρόνου και ίσως έχοντας την δυνατότητα για εκείνα τα σημεία που πρέπει να εξεταστούν με τον Αντιπρόεδρο κύριο Κάλλας, γι' αυτό ε, συνάδελφοι θα ήθελα να προτείνω να συνεχίσουμε αμέσως και παρακαλώ όποιος θέλει να αποχωρήσει, να αποχωρήσει ήσυχα και ήρεμα. Και τώρα μπορούμε να επισπεύσουμε το σημείο 6. Αυτή θα ήταν η πρότασή μου. Το λέω στα αγγλικά η ειδική έκθεση 11 ε, του 2008 του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ε, διαχείριση για την ε, αποθήκευση δημητριακών. Ο Γιάν Μούλτερ είναι το αρμόδιο μέλος για αυτό το θέμα. Χαιρετίζω από το Ελεγκτικό Συνέδριο τον κύριο Άλλα Νίση λέει. Και θα δώσουμε τον λόγο τώρα ο κύριος Μούλτερ. Ο κύριος εισηγητής λοιπόν θα έχει τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Παρεμβαίνω Πιστεύω βέβαια ότι πρέπει να παρέμβει και το ελεκτικό συνέδριο και σε σχέση με την δική μας συνάντηση στο Ευρωκοινοβούλιο πρέπει στις 5 να παρέμβω, πρέπει να ε, βιαστώ λοιπόν για να τα καταφέρω. Χαίρομαι λοιπόν που μπορώ να κάνω κάτι ε, αυτό το απόγευμα και να ανακουφίσω τη... για αυτό το θέμα γιατί έχουμε μια έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου που είναι θα έλεγα θετική πρόκειται για την δημόσια αποθήκευση σιτηρών μητριακών. Ξέρω ότι και ο κύριος Ιτον Χάρης είναι, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για αυτό το θέμα και η γενική έκθεση είναι θα έλεγα αισιόδοξη και συμμερίζομαι αυτά τα συμπεράσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω με καλό τρόπο διαχειρίζεται αυτή την, ε, αυτό το θέμα. Όπως σε όλες τις περιπτώσεις μπορούν να υπάρξουν και εδώ βελτιώσεις. Οι βελτιώσεις θα εξεταστούν από το, αξιολογηθούν από το ελεγκτικό συνέδριο. Γενικά συμφωνώ με, τις, ε, με τα συμπεράσματα του ελεγκτικού συνεδρίου. Συμπεράσματα είναι ότι θα πρέπει να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι καλύτεροι τρόποι ε, της ε, μείωσης και αντιμετώπισης των γραφειοκρατικών δράσεων, να λαμβάνουμε υπόψη τις ε, τιμές αγοράς, τις τιμές εξαγωγών και να βρούμε άλλες δυνατότητες. Στην έκθεση δίνει, δίνεται μια, ένα παράδειγμα και για τη βιοεθανόλη θα πρέπει να ε, δούμε αυτό το θέμα. Ως πιλωτικό πρόγραμμα θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι συμβαίνει αυτό. Όπως λοιπόν με, όλες, ε, με όλους τους ελέγχους ε, θα πρέπει να γίνεται ένας υπολογισμός Ποιε είναι, ποιες είναι οι δαπάνες, το κόστος των επιθεωρήσεων και ποια είναι τα ωφέλη και η αξία που παρέχεται. Και υπογραμμίζοντας κάτι το οποίο δεν βρίσκεται στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, αυτό είναι το ότι κάνουμε λόγο για την παρέμβαση. Είναι κάτι το οποίο είναι αναγκαίο <clears throat> για την ίδια την αγορά και θα είναι αναγκαίο επίσης και ως στρατηγικό εργαλείο πέρα από το πλαίσιο αγοράς σε περιόδους ε, ενεργειακής πανίδας ε, και ε, θα είναι σημαντικό νομίζω η αποθήκευση σιτηρών να προβλέπεται για περιόδους κρίσεως στο μέλλον. Δεν χρειάζεται κανείς να διαβάσει τη βίβλο για να δει κανείς τις περιόδους ισχνών Ελλάδων. Ε, είναι χρήσιμη η αποθήκευση λοιπόν για την αντιμετώπιση ε, τέτοιων ε, προβλημάτων. Ζητώ συγγνώμη από όλους. Πρέπει να αποχωρήσω. Θα μείνω για πέντε λεπτά. Πρέπει να πάω σε άλλη αίθουσα. Ζητώ συγγνώμη για αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ για την κατανόηση. Σας ευχαριστούμε και έτσι λοιπόν περνάμε αμέσως στον κύριο Άλλα Νίσιλε του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Έχετε τον λόγο παρακαλώ. Uh, Σας ευχαριστώ, ε, μέλη της, Επιτροπής Ελέγχου Προεκολισμών. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μούλτερ για τα θετικά σχόλια που έκανε για τις συστάσεις όσον αφορά το έγγραφο εργασίας και την ευθυγράμμιση με τις δικές μας συστάσεις. Και τώρα κάποια σχόλια σύντομα για την ε, έκθεσή μας όσον αφορά την ε, διαχείριση για την ε, αποθήκευση εισιτήρων. Αποφάσισε το ελληνικό συνέδριο να κάνει αυτούς τους ελέγχους το 2007 σε μια κατάσταση όπου τα αποθέματα σιτήρων είχαν φτάσει σε υψηλά επίπεδα, κυρίως λόγω της διεύρυνσης του 2004. Έκτοτε η κατάσταση άλλαξε βέβαια αυτή τη στιγμή δεν έχει σημαντικά αποθέματα σιτηρών η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πρόσφατη πτώση ε, των τιμών ε, σε κάποια κράτη-μέλη ε, οδήγησε σε αυτή την τάση. Τώρα αυτό που κάναμε σε σχέση με την αποθήκευση σιτηρών και ιδιαίτερα με την ελαχιστοποίηση του κόστους και την μέγιστοποίηση των εσόδων αξιολογήσεις ε, και η ε, στάθμιση της καλής χρηστής διαχείρισης μέσω της ε, διαδικασίας αποθήκευσης διασφαλίζεται ότι το κόστος θα ελαχιστοποιείται, θα βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα. Αυτό που βρήκαμε από πλευράς των ελέγχων και οι απαντήσεις σε κάποιες σχετικές χρήσιμες παρατηρήσεις και σχόλια. Η έκθεση βρίσκει ότι γενικά η διαχείριση ε, των δράσεων για την αποθήκευση και οι διαδικασίε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν συνολικά ικανοποιητικές και ικανοποιητικά. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα στα οποία μπορούν να σημειωθούν βελτιώσεις, ιδιαίτερα οι διεργασίες ε, για τη διάθεση που δεν διασφαλίζουν πάντα ότι το καθαρό κόστος ε, της παρέμβασης θα ελαχιστοποιείται ή ότι δεν θα παραμένουν αυτά τα, ε, αυτοί οι όγκοι στην αποθήκευση, σε καθεστώς αποθήκευσης πέρα από ό,τι αναγκαίο. Και ιδιαίτερα όσον αφορά την, ε, την υψηλή, υψηλότερη αξία που θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω εξαγωγών. Έλλειψη ευελιξίας με αποτέλεσμα κάποια αποθέματα να παραμένουν μεγαλύτερο χρόνο σε αποθήκευση αποθήκευση ε, πράγμα το οποίο οδηγεί σε αύξηση κόστους και εδώ και η ποιότητα και η τοποθεσία ε, δεν ε, λαμβανόντουσαν πάντα υπόψη δεύτερον επιστροφές κονδυλίων στα κρατημέλη που μπορεί να υπερβαίνουν το κόστος που έχει προκληθεί πράγμα το οποίο οδηγεί σε υπερβολική θα έλεγα αντιστάθμιση και τρίτον, η αποθήκευση και από του κονδυλίου και οι δραστηριότητες που δεν συσχετίζονται άμεσα στις παρεμβάσεις για αποθήκευση. Αυτό συνέβαινε με την διάθεση ε, για τιμές χαμηλότερες από τις τιμές αγοράς ε, για την βιοεθανόλη και τον ε, βιομηχανικό αυτοκλάδο. Αυτό έχει επιπτώσει στη διαφάνεια του, των λογαριασμών του ε, προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνιστά λοιπόν το ελεγκτικό συνέδριο ότι τα εξή στοιχεία θα πρέπει να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη αξιολογώντας και αποτιμώντας ε, την διάθεση ποιότητα και τοποθέτηση ε, σημείο γεωγραφικό ε, αποθήκευσης αυτού του προϊόντος βλέποντας, προσέχοντας ε, την υψηλότερη προσφορά που μπορεί να επιτευχθεί ε, για τη διάθεση ή και την χαμηλότερη τιμή που μπορεί να απαιτείται για εξαγωγή. Συνιστά επίσης το συνέδριο για να βελτιωθεί η δημοσιονομική διεργασία το κόστος των δραστηριοτήτων που δεν συσχετίζονται άμεσα με την αποθήκευση των σιτηρών να μην επιβαρύνει τις ε, ε, δράσεις αυτές όσον αφορά επίσης και τις δραστηριότητες στον τομέα της βιοεθανόλης πρέπει να υπάρχει ένα διαφανέστερο πλαίσιο και να υπάρχει η δυνατότητα αντιστάθμισης όσον αφορά τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να αναθεωρηθούν λοιπόν οι διεργασίες από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι υπολογισμοί για την επιστροφή, για την ε, κάλυψη των, ε, του κόστους ε, σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Αυτό μπορεί να έχει σημαντική επίπτωση αν αυξηθούν τα αποθέματα θέματα σιτηρών στο μέλλον. Συνιστά έντονα το Συμβούλιο να υιοθετηθούν αυτές οι βελτιώσεις των δυνατών ταχύτερων. Και κατά τη διάρκεια των ε, διακριβώσεων αυτών και τα κυριότερα συμπεράσματα που ε, συμφωνήθηκαν όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην ενδιάμεση αναθεώρηση της ΚΑΠ δεν αμφισβητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την σκοπιμότητα της αποθήκευσης σιτηρών. Οι προτάσεις ε, συνεπάγονται στο να διατηρηθεί η ε, κρατική παρέμβαση ώστε να υπάρξει ένα δίκτυο ασφαλείας. Και να μην ε, υπάρξει αρνητική επίπτωση μεσοπρόθεσμα στην ε, δραστηριότητα ε, αποθήκευσης. Συνολικά κύριε Πρόεδρε η έκθεση μπορεί να φαίνεται υπερβολικά τεχνική στον αναγνωστή όμως εμπεριέχει χρήσιμες και επικοδομητικές συστάσεις και σχετικά εύκολο θα ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εισαγάγει και να υιοθετήσει αυτές τις συστάσεις σε αυτή τη συγκυρία χαμηλών αποθεμάτων και να διασφαλιστούν έτσι τα θετικά αποτελέσματα των συστάσεων τον Ευχαριστώ Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε για την εισαγωγή σας. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει κάποια παρατήρηση. Ίσως η Επιτροπή πρώτα λοιπόν, παρακαλώ. Με Ο ε, για τα Γεωργία. δεν ήξερα ότι θα αυτή τη μερισία διάταξη, δεν είναι προφτασε να έρθει. Θα σας δώσω μόνο μια πρώτη αντίδραση εγώ. Χαιρετίζουμε τις θετικέ παρατηρήσεις ε, του ηλεκτρικού συνεδρίου στον αφορά το σύστημα αυτοποθήκευσης δημητριακών. Ε, χαιρετίζουμε τις συστάσεις που υποβάλλουν για τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης. Δεν συμφωνούμε με όλα, αλλά οπωσδήποτε εκτιμούμε την επικοδομητική προσέγγιση του συνεδρίου. Αυτή τη στιγμή το ποσοστά είναι στην τάξη του 0 ε, ε, πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Οπωσδήποτε θα εξετάσουμε τις συστάσεις και θα δούμε πώς θα δυναμώσουμε το ρόλο σαν μια εξασφάλιση ε, έναντι υπερβολικά χαμηλών τιμών. Σημειώνουμε λοιπόν αυτά παρόλο που αυτή η στιγμή δεν είναι απαραίτητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μούλη για το έγγραφο του, να απαντήσουμε σε κάποιες παρατηρήσεις που έγιναν. Όσον με το σύστημα των διαγωνισμών πάντα είχαμε κάτι τέτοιο, πάντα είχαμε δημοπρατήσεις και μέσα στα πλαίσια του διάμεσου ελέγχου, του health check, πρόκειται να τροποποιηθεί το σύστημα, αλλά δεν είναι ακόμα λειτουργική η τροποποίηση αυτή. Όσον αφορά τις προσπάθειες ε, περαιτέρω εκλεπτισμού του συστήματος που χρησιμοποιούμε για την επιστροφή του κόστους, όταν ε, συζητάτε μάλιστα δύο πωλήσει και αγορές ε, το συνέδριο λέει ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε πού αγοράστηκε το προϊόν, πού βρίσκεται κλπ. Αυτό βέβαια θα περίπληκε ακόμη περισσότερο μια ήδη περίπλοκη κατάσταση. Θα ήταν καλύτερο να αφήσουμε ε, το θέμα αυτό να οργανωθεί από τα κράτη-μέλη. Πρέπει να έχετε βρώμη με υψηλό ποσοστό πρωτεΐνης, αυτό είναι πολύ καλό για ζωοτροφές. Δεν το χρησιμοποιήσετε εκεί για ε, ζωοτροφές. Αν θέλετε το χρησιμοποιήσετε όμως για ε, μπύρα, για την παραγωγή μπύρας, θα ήταν αιτική η περιεκτικότητα αυτής της πρωτεΐνης. Πρέπει λοιπόν να κρίνει κανένας σωστά. Πώς θα δοθούν κίνητρα στα κράτη-μέλη για να μειωθεί το κόστος. Αυτή τη στιγμή χαιρόμαστε ότι επιστρέφουμε κάποια χαμηλότερα ποσά από ό,τι είχε προβλεφθεί. Εμείς προσπαθούμε να κλείσουμε τα θεωρητικά κενά που βρήκε όμως το ηλεκτρικό συνέδριο. Στη θεωρία μόνο, στην πράξη δεν έχουμε το πρόβλημα. ζητήσετε από την Κομισιόν να δώσει περισσότερα κίνητρα στη κράτη-μέλη για να καταστήσει πιο ειδονική τη στιγμή πώλησης του προϊόντος ή μα ζητάτε να ελέγχουμε καλύτερα τι ημερομηνίε προς προ τα Μέλη. Εμεί ελέγχουμε ει βάθο τι ε, διοικητικέ αυτέ διαδικασίε. Ξέρω ότι είναι μακρά η διαδικασία, γιατί καμιά φορά δεν πιστεύουμε τα στοιχεία που μας στέλνουν και έχουμε μακρές ζητήσει με τα κράτη-μέλη πριν να ικανοποιηθούμε ότι τα στοιχεία που μας στείλαν ήταν σωστά και τότε ορίζουμε το κόστος που πρέπει να ε, επιστραφεί. Ε, καμιά φορά χρειάζεται να πάει κανένας επιτόπου βέβαια για να ελέγξει. Θεωρούμε, χωρίς να πούμε σε λεπτομέρειες, ότι η μέθοδος ε, υπολογισμού του της ποσότητας εισόδου των αποθεμάτων αυτών χωρίς δηλαδή πραγματικές ε, κινήσεις είναι υπερβολικά ε, γενναιόδρας από τα κράτη-μέλη. Εμείς προσπαθούμε τώρα να βελτιώσουμε τη μεθοδολογία αυτή υπολογισμού. Γιατί έχουμε κάποιες ποσότητες που εντάσσονται μέσα στα αποθέματα που δυσκολεύουν όλη την κατάσταση. Ο κ. Μούλτερ χρειάστηκε βέβαια να φύγει όπω μα είπε, αλλά εκείνο είχε προτείνει να δημιουργήσουμε ένα απόθεμα ασφάλειας. Αυτό δεν ήταν κάτι που ουσίασε νομίζω το ελληνικό συνέδριο, ήταν η ιδέα του κυρίου Μούλτερ, οπωσδήποτε στο διάμεσο έλεγχο, στην health check αυτό, το Συμβούλιο είπε ότι θα πρέπει να παραμείνει η ε, παρέμβαση σαν ένα μέσο ε, εξασφάλισης αν θέλετε. Αυτό θα ήταν σημαντικό αν υπήρχε ξαφνικά μια ξηρασία Φερρυπίν. Και χρειαζόταν να χορηγήσουμε επιστηστική βοήθεια. Αυτό είναι βέβαια ένα θέμα της έγκαιρης πρόβλεψης των εξελίξεων μάλλον και όχι να έχουμε τεράστιες ποσότητες δημητριακών που να βρίσκονται αποθηκευμένα εδώ και εκεί. Αυτά πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Ο κύριος Σοντή. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Μούλτερ για τη σημαντική του εργασία και θα ήθελα να υποβάλω και μια ερώτηση που είχα υποβάλει και στο παρελθόν. Ποιο είναι το καθεστώς του εγγράφου αυτού. Στην σελίδα 6 λέγεται ότι είναι μία σύσταση της ε, Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού για να ενταχθεί μέσα στην έκθεση του εισηγητή. Εγώ είμαι εισηγητής όμως, αυτό δεν έχουμε ψηφίσει αυτό το κείμενο. Τι είναι αυτό, είναι πρώτος κ. Μούλτερ, τι είναι. Äh, αυτό κατά βάση είναι ένα έγγραφο εργασίας με διάφορες συστάσεις, με διάφορα συμπεράσματα. Εσείς είστε το γενικό συγγητής. Ε, δική σας απόφαση θα είναι τι θα εντάξει από όλα αυτά μέσα στα πλαίσια της απαλλαγής για το 2007 και τι όχι. Αυτό είναι το καθεστώς του εγγράφου. Εντάξει. Άλλος που θα ήθελε το λόγο πάνω στο σημείο αυτό. Όχι. Ο συγητής ε, η Κομισιόν μίλησε. Εντάξει, μπορούμε να κλείσουμε το σημείο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και περνάμε στο επόμενο σημείο. Το σημείο 15 που είχαμε πει θα εξετάσουμε τώρα. Προ μια διοργανική συμφωνία σχετικά με την έννοια του αποδεκτικού κινδύνου σφάλματο στα κοινοτικά προγράμματα. Θα ήθελα να χαιρετήσω εδώ τον Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Σιμ και θα ήθελα αμέσω να του δώσω και το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, εξότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε αρκετά χαρούμενοι. Διότι δύο με τρία χρόνια προσπαθειών παρήγαγαν ένα πραγματικό έγγραφο το οποίο μπορεί να είναι σημαντικό βήμα προόδου για να βελτιώσουμε την αρχιτεκτονική του ελέγχου. Είμαι πολύ χαρούμενος που προσεκλήθη να σας παρουσιάσω την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου. Σύντομη και σαφή είναι η ανακοίνωση, ελπίζω να απολαύσατε την αναγνωσή της. Σήμερα δεν θα επισέλθω σε τεχνικές λεπτομέρειες, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε παρά τον προφανή κίνδυνο να παρεξηγηθούμε. Η πιθανότητα παρεξηγήσεως των προθέσεών μας λόγω της ανακοινώσεως είναι πάρα πολύ μεγάλη και γι' αυτό θα ήθελα να αναφέρω κάποια σημεία. Περί τίνος δεν πρόκειται αυτή η πρωτοβουλία. Τι δεν θέλει να κάνει. Δεν θέλουμε να καθορίσουμε ένα αποδεκτό επίπεδο απάτης. Δεν υπάρχει ανεκτό επίπεδο απάτης. Μηδενική ανοχή είναι η πολιτική που ακολουθούμε για την απάτη. Είναι αυστηρή συνέχεια αυτή η πολιτική μας αυστηρή παρακολούθηση κάθε ατασταλίας που διαπιστώνουμε εμείς ή το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Όπως σας πει κύριε Χίμπνερ αύριο, τα ποσά που ανακτώνται αυξάνονται. Ανεκτός κίνδυνος δεν αφορά ήπια προσέγγιση επισφαλμάτων, αλλά θέλουμε εκ των προτέρων συμφωνία διαφανή για το επίπεδο σφαλμάτων που θα θεωρηθούν τόσο σημαντικά που αμφισβητούν το σύστημα. Και δεν δίνεται θετική δήλωση αξιοπιστίας και κινδυνεύει ε, η απαλλαγή. Και θα πρέπει να σταματήσει η χρηματοδότηση κάποιων τομέων ή να επαναξεταστούν οι κανόνες. Αποδεκτός κίνδυνος καθορίζει τα όρια μεταξύ σφαλμάτων προς διόρθωση και συστηματικών, συστημικών αδυναμιών που αμφισβητούν γενικότερο σύστημα. Δεύτερον, δεν είναι δικαιολογία για να μην δοθεί θετική δήλωση εξοπιστίας φέτος. Όπως είπα, υπομίζομαι τις ευθύνες για τα επιτευθέντα αποτελέσματα και είμαι υπερήφανος για την επιτευθύσα πρόοδο. Τον Φεβρουάριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υιοθετήσει την πρώτη έκθεση συνεπιών για τον οδικό χάρτη προς θετική δήλωση εξοπιστίας και υπάρχουν πάρα πολλές βελτιώσεις παρά τα όσα αντικατοπτρίζονται στα ποσοστά σφάλματος που στο ελεκτικό συνέδριο. Αυτό δεν αντικαθιστά βελτιώσει μελλοντικέ όσον αφορά βέβαια τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Οι προσπάθειε για την βελτίωση πρέπει να συνεχιστούν. Σαν ένα μέρο των όσων παρουσιάζω σήμερα, υπάρχει και η ανάγκη βελτίωση. Τονίζεται επανειλημμένα η ανάγκη βελτίωση. Όσον αφορά τα ιδιωτικά ταμεία, λέμε ότι το 11% σφαλμάτων θα πρέπει να μειωθεί έτσι περαιτέρω, που είναι το ελάχιστο επίπεδο, βάσει των ελέγχων. Εφαρμόζοντα καλύτερα του θεσπιστέτε κανόνε, διοικητικέ δαπάνε στον τομέα μου, ίσω οι υπολογισμοί μα οδηγήσουν σε ανεκτό επίπεδο κινδύνου που είναι κάτω από το 2%. Τέταρτον, δεν προσπαθούμε να εκβιάσουμε κανέναν ώστε να μας δώσει περισσότερους πόρους για τους ελέγχους. Από τις πρώτες συζητήσεις μας με τα κράτη-μέλη γνωρίζουμε ότι κάποια από αυτά ανησυχούν τα μάλα για αυτά τα προβλήματα και υποψιάζονται ότι είναι κρυμμένη η έκκληση για περισσότερους ελέγχους και περισσότερες θα πάνε σε τα κράτη-μέλη. Αυτή η ανακοίνωσή μας. Όπως βλέπετε στο κείμενο είμαστε αρκετά πραγματιστές. Όσον αφορά τα θετικά ταμεία ίσως να εξεπλάγεται διαβάζοντας τα κράτη-μέλη λένε ότι το κόστος ελέγχου είναι 0,7% των συνολικών δημοσίων δαπανών για τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη Επενδύσεων. Και το σημείο ε, ισορροπίας για αποτελεσματικούς ελέγχους είναι περίπου στο επίπεδο σφαλμάτων το 4%. Για να το πετύχουμε αυτό όμως χρειαζόμαστε άλλα 680 εκατομμύρια για το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο. Είναι ρεαλιστικό να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να μας δώσουν ε, παραπάνω χρήματα και καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες. Πέμπτον, το επίπεδο ανεκτού κινδύνου δεν είναι μια παραχώρηση ούτε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε για τα κράτη-μέλη. Κανείς δεν θέλει να μας απαλλάξει από τις προσπάθειες βελτιώσεως της διαχείρισης όλα τα επίπεδα. Ανταυτού, ο ανεκτός κίνδυνος αφορά την χρήση των σωστών εργασ... εργαλείων για το σωστό στόχο. Δηλαδή, σωστό δόλωμα και σωστό ψάρι και αν πιάσει το ψάρι μην τα αφήσει φύγει αν συμφωνήσει η νομοθετική αρχή για το ελάχιστο επίπεδο κινδύνου, θα πρέπει τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμορφωθούν. Δεν επικρίνουμε το ελεκτικό συνέδριο με αυτά που θα πούμε τώρα, ούτε την τρέχουσα μεθοδολογία του ελεκτικού συνεδρίου, αλλά θα πούμε ότι ανεκτό κινδύνο ήταν η ιδέα του ελεκτικού συνεδρίου στην αρχή και προτάθηκε το 2004. Θα, θέλουμε να... θα θέλετε να ακούσετε τι έχει να πει το ελεκτικό συνέδριο άμεσα. Απλώ ήθελα να πω ποιο είναι ο πνευματικό πατέρα τη ιδέα. Να στραφώ τώρα προς την ε, πρόταση της ανακοινώσεως. Στην ανακοίνωση σας δίνουμε ε, ένα μοντέλο. Διερευνούμε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των ποσών που δαπανώνται για τους ελέγχους και το επίπεδο σφαλμάτων που εντοπίζεται από τους ελέγχους. Εκτιμούμε ότι το κόστος συμπληρωματικών ελέγχων και συγκρίνουμε αυτό με τις οικονομικές συνέπειες που έχει το σφάλμα ε, που θα μπορούσε να αποφευθεί ενδεχομένως. Είναι αρκετά εύκολο αυτό και έχουμε παρουσιάσει τα πλέον απλά μοντέλα. Χρησιμοποιώντας αυτό το μοντέλο σε δύο παραδείγματα υπολογίσαμε το σημείο εξουδετερώσεως του κόστους. Εκεί βλέπουμε θεωρητικά τι πρέπει να δαπανούμε για τους ελέγχους και ποιο επίπεδο ελέγχου πρέπει να γίνεται αποδεκτό. Αυτό όμως δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Θα ήθελα να τονίσω ότι ενώ μια οικονομική τέτοια ανάλυση είναι σημαντική για να κατανοήσουμε τα επίπεδα του ελέγχου. Καθορισμό ανεκτού επίπεδου σφαλμάτων είναι πολιτική απόφαση. Ανθρωπιστική βοήθεια, φερειπίνει, είναι όπου χαμηλό κόστο ελέγχου μπορεί να είναι αποδεκτό, ούτω ώστε να δοθεί η βοήθεια γρήγορα. Όμω, άλλου τομεί που υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την εικόνα προβάλλεται και υπάρχουν πολιτικέ στοιχείε να ληφθούν υπόψη, ίσω το κόστο είναι περισσότερο βαρύ, περισσότερο η πολιτική απόφαση από το κόστο για κάποιο συγκεκριμένο τομέα, αν θεωρηθεί ότι ο υπολογισμό δίνει ένα σημείο εξισορρόπηση σε πολύ μη ρεαλιστικά επίπεδα, με πάρα πολλέ δαπάνε για τον έλεγχο, έχει τρει επιλογέ. Είτε αρνείσαι την αδειοδότηση αυτών των μεγαλύτερων δαπανών για τον έλεγχο, να αντιταχθεί στη δαπάνη και μπορεί να δεχτεί και επίπεδο κινδύνου και αν υπάρχει μεγάλος κινδύνος, ίσως περικόπτει στις δαπάνες στον τομέα. Ίσως απλουστεύει στην εξίσωση. Απλούστευση. Κανόνες επιλεξιμότητας είναι περίπλοκοι σε κάποιους τομεί. και δημιουργούν σφάλματα. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε όσου κανόνε επιλεξιμότητα για απλούστευση. Δεν υπάρχει κόστο αν δεν υπάρχουν κανόνε και δεν υπάρχουν σφάλματα. Αν θέλουμε να πετύχουμε συγκεκριμένου στόχου πολιτική, πρέπει να καθορίσουμε κανόνε επιλεξιμότητα. Δεόντω, η ανάπτυξη τη υπαίθρου είναι ένα παράδειγμα. Απλουστεύοντα και βγάζοντα λεπτομερή κριτήρια επιλεξιμότητα, θα βγάζαμε και τι θετικέ συνέπειε για το περιβάλλον. Και είναι και θέμα χρονικού συντονισμού Υπερβολική απλούστευση σημαίνει επανεξέταση βασικών πράξεων που είναι κάτι χρονοβόρο. Αν συμφωνηθούν τέτοια μέτρα, τα ανεκτά επίπεδα κινδύνου θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Εν τω μεταξύ, πρέπει να κινηθούμε βάσει των υφισταμένων κανόνων. Γενικά, οι πολίτες της Ευρώπης περιμένουν να συμφωνήσουμε με πολιτικών και να πετύχουμε αποτελέσματα. Πολιτικές επιταγές πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και όπως λέει και το ελεκτικό συνέδριο, ο τρόπος διανομής των κοινοτικών πόρων σε εκατομμύρια δικαιούχους βασίζονται σε ατομικές δηλώσεις εκείνων που δέχονται τους πόρους. Αυτό βέβαια εκεί ελοχεύουν κίνδυνοι. Σαν νομοθέτες καταλαβαίνετε ότι κάποια, κάποιοι μηχανισμοί είναι εγγενώς ε, παρακινδυνευμένοι και εμείς θα πρέπει να αξιολογήσουμε τους κινδύνους. Δεχόμενοι κάποια σφάλματα που θα διορθώνονται μετά από εντοπισμό. Η ανακοίνωση λοιπόν δεν το κάνει αυτό για σας. Η δουλειά των νομοθετών είναι απαραίτητη. Η ανακοίνωση σας παρουσιάζει μια προσέγγιση. Σας δίνει μια βάση για τη λήψη των αποφάσεών σας. Αυτό δημιουργεί στέρεη βάση για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαι πεπισμένος ότι η συζήτηση για το ανεκτό επίπεδο κινδύνου και σφάλματος αξίζει τον κόπο για όλους μας. Πρέπει να συζητηθεί. Χρειάζεται διοργανική συζήτηση με Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ελεκτικό Συνέδριο βάσει της παρούσης ανακοινώσεως. Εάν τα συμπεράσματα της συζητήσεως θα είναι θετικά, Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβεί σε περαιτέρω ανάλυση του ανεκτού κινδύνου, κυρίως για την έρευνα, την ενέργεια, τις μεταφορές, εξωτερική βοήθεια, ανάπτυξη, διεύρυνση και διοικητικές δαπάνες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Περιμένω πώς και πώς να ακούσω τα σχόλιά σας και τη διεξαγωγή της συζητήσεως. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Το λόγο έχει ο εισηγητής μας κύριε Σοντή, αν θέλει να κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Μάλιστα, πρόεδρε. Δεν ήξερα ότι ήμουν εισηγητής. Μα είσαστε για τα πάντα εισηγητής, κύριε Οντή, φέτος. Ε, εγώ θετικά το βλέπω. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Καλάς για το έγγραφο αυτό θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο και εσείς ο ίδιος Πρόεδρε ε, ήσασταν από εκείν, τους προκαταγωνιστές ε, για την εντύπωση του ε, προγράμματος αυτού και βλέπω ότι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να εξετάσουμε. Θα είμαι αρκετά σύντομος γιατί έχω μια σκέψη που με απασχολεί και το λέω ειλικρινά προς τον κύριο Αντιπρόεδρο και προς το ηλεκτρικό συνέδριο. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο ορισμός του ε, επίπεδου αποδεκτού σφάλματος ε, είναι πολιτική απόφαση. Λέμε πάντα ότι πρέπει να σεβόμαστε τους διεθνούς κανόνες ελέγχου. Αυτό πρέπει να μπορεί να ελέγχεται σε εθνικό επίπεδο, γιατί στους διεθνούς κανόνες ο ελεγκτής είναι εκείνος που αξιολογεί το κίνδυνο. Άμα δούμε τις εκθέσεις του ελεκτικού συνεδρίου, όχι εκεί που αναφέρονται τα συμπεράσματα, αλλά όσον αφορά την ευθύνη του ελεκτού, που υπάρχει μια παράγραφος 4, που λίγο πολύ αντικατοπτρίζει τους διεθνούς κανόνες και λέγεται η επιλογή της διαδικασίας εξαρτάται από την κρίση του ελεκτού, που εξετάζει επίσης το αποδεκτό κίνδυνο, πρωτοβουλίε κλπ. Και ο ελεγκτής είναι εκείνο ο οποίος αξιολογεί τον κίνδυνο γενικά και τον αποδεκτό κίνδυνο γενικά. Και να η πολιτική είναι εκείνη που θα ορίσει αυτά τα επίπεδα. Η πολιτική προσφανώς θα χρηματοδοτήσει και οι φορολογούμενοι παρατηρούν προσεκτικά, δεν μπορούν να χρηματοδοτούν τα πάντα στον αφορά το κόστος ελέγχου θα έπρεπε η να έχουμε από το συλλεκτικό συνέδριο κάποια σωστή ε, εξασφαλίσεις όσον αφορά τους οργανισμούς αυτούς κλπ. Και βου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ορίσει ένα επίπεδο κινδύνου για τις δικές της υπηρεσίες, για εκείνες τις υπηρεσίες δηλαδή τις οποίες ελέγχει. Αλλά δεν ξέρω, αυτό είναι μια ιδέα που ρίχνω εδώ πάνω στο τραπέζι. Θα με ενδιαφέρει να ακούσω τις απόψεις που έχετε να μου παρουσιάσετε σχετικά. Πρώτος, ευχαριστώ. Είναι πολύ καλή εισαγωγή νομίζω για το ελεκτικό συνέδριο. Κύριος Μπονίτσι, έχει να μας πει κάτι. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πρόεδρε. Το ελεκτικό συνέδριο αυτή τη στιγμή εξετάζει την ανακοίνωσή του. Δεν έχω λοιπόν μια θέση του συνεδρίου ακόμα. Μπορώ να σας δώσω κάποιες απόψεις σε προσωπική βάση για την ανακοίνωση αυτή. Καταρχήν θεωρώ ότι η συζητήση στην ανακοίνωση ασχολείται με το οικονομικό βέλτιστο όπως λέμε. Ένα οικονομικό βέλτιστο δεν είναι απαραίτητα ένα, ε, σε ένα επαρκές επίπεδο κινδύνου, αλλά να λάβει υπόψη το τι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η απόψη μας από μερικά χρόνια που δημοσιεύτηκε είχαμε πει ότι είναι θέμα των πολιτικών αρχών να το μελετήσουν όχι εμείς δεν πρέπει εμείς να το καθορίσουμε Παρακολουθούμε λοιπόν προσεκτικά και με ενδιαφέρον τη συζήτηση. Υπάρχουν ήδη κάποια αποτελέσματα. Σημαντικά, ενδιαφέροντα. Εγώ παραδείγματος χάρη εξεπλάγει από το κόστος ελέγχου σε ιδιωτικό ταμείο 0,7-0,8% πριν από κανένα δύο χρόνια ήταν της τάξης του 3% νομίζω Αυτή είναι η εντύπωση, όχι βάσει τη δική μα εργασία, αλλά αυτά που είχε πει η Κομισιόν. Και νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία ήταν πιο ακριβή. Αλλά κοιτάζοντα τη Γεωργία, βλέπατε ότι το κόστο λέγουν τη τάξη του 4%. Και μετά κοιτάτε τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα στη Γεωργία είναι βέβαια ανώτερα από τα αποτελέσματα στα κατά μία που είναι πολύ προβληματικά. Και γι' αυτό η άμεση μου απάντηση θα ήταν ότι πράγματι πρέπει να γίνουν περισσότερα στο τομέα των ερωτικών ταμείων. Και αυτή είναι μια θέση που εξέφρασα στο παρελθόν στη δική σας επιτροπή, ήδη όταν συζητούσα τις εκθέσεις του Γενικού Διευθυντή. Διαβάζοντας βλέπει κανένα ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στη διαχείριση του τομέα. Πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα. Τώρα κατά πόσον πρόκειται για το ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων που ισχύουν αυτή τη στιγμή ότι θα πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι. Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Όσον αφορά την περιβαλλοντική πλευρά της Γεωργίας, έχουμε ακριβώ την αντίθετη κατάσταση. Το κόστος του ελέγχου είναι στις τάξεις 13%. Μας φαίνεται υπερβολικά υψηλό, λόγω των αποτελεσμάτων που έχουμε δώσει στο τομέα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να αναλυθούμε κατά πόσο η έννοια αυτή είναι αντιστική και χρήσιμη για να πετύχουμε το απαραίτητο και εύκολο αποτέλεσμα. Αυτά είναι κάποια στοιχεία εδώ που μπορώ να σας δώσω. Μετά θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να πετύχουμε αυτό το οικονομικό ε, ε, βέλτιστο. Γιατί αυτό είναι κάτι που υπάρχει σε διάφορες γραμμικές παροστάσεις ε, της Κομισιόν κλπ. Πρόκειται για την ε, ε, αξιολόγηση του κόστου ελέγχου βάσει του κόστους λειτουργίας. Ο κύριος Κάλλας είπε ότι υπάρχει εδώ συνένεση, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε άλλους τομείς. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε πριν να φτάσουμε εκεί. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ενδυναμώσουμε τη βάση πληροφορίας για τους δύο τομείς που εξετάστηκαν. Δηλαδή υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα και θα πρέπει να έχουμε αρκετά στεναρό αποτέλεσμα, αρκετή εμπιστοσύνη, το ώστε να ξέρουμε ότι τα ποσά που αναφέρονται είναι τα σωστά για να μπορέσουμε να βασιστούμε σε αποφάσει μα. Προηγουμένω, με ρωτάγατε, ξαναρωτάγατε, αυτά τα 150 σημεία α, ήταν ένα σωστό δείγμα του συνόλου ή όχι. Εδώ έχουμε κάτι που είναι πολύ πιο κρίσιμο, χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες. Και είναι καλό να συγκεντρώσει προσοχή της Κομισιόν εδώ. Αν κάποιος θέλει να σωστά κάποιους πόρους και κάποια ταμεία, χρειάζεται πληροφορίες για το πόσο αποτελεσματική είναι η έλεγχη και το πόσο κοστίζουν οι έλεγχοι και ποιες είναι οι επιπτώσεις των ελέγχων αυτών. Αυτό συζητάμε. Είναι πολύ καλό λοιπόν το σημείο κίνησης εδώ. Και είναι σημαντικό για το σύνολο της συζήτησης εδώ. Παρ' όλα αυτά θα έλεγα ότι χρειάζεται μια ευρύτερη βάση δεδομένων. Μπορεί να μας πει κανένα. ναι, αλλά έχουμε όμως προβλήματα με τις προφορές από τα κράτη-μέλη, δεν υπάρχει κλπ. κλπ. Όλα αυτά ίσως είναι αληθή. Υπάρχει ένα πρόβλημα στον τομέα. Αλλά δεν είναι αυτή εδώ η μόνη πηγή πληροφοριών. Ίσως θα πρέπει να ελέγξουμε περισσότερο μέσω κάποιων ελέγχων της δειγματοληψίας για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αυξήσουμε ε, την βασιμότητα. Αν δεν έχουμε αυτές τις πληροφορίες, είναι κάπως προβληματικό θα έλεγα να εξετάσουμε το θέμα του αποδεικτού κινδύνου σφάλματος. Γιατί ή τα αφήνουμε όλα ελεύθερα ή στο άλλο άκρο όλα ελέγχονται και θα πρέπει να γίνουν οι υπολογισμοί ανάμεσα στις διευθυντές. Τέλος πάντων αυτή που σας παρουσίασα ήταν μια προσωπική μου άποψη. Και διαβάζω στο έγγραφο σας είπα ότι θεωρώ είναι καλό που η Κομισιόν εξετάζει αυτό το τομέα. Από την άλλη μεριά θεωρώ ότι θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να υπάρχει μεγαλύτερη ακρίβεια στις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για να εξεταστεί το γενικό θέμα του αποδεκτού σφάλματος. Είναι πιο ευρύ αυτό. Το οικονομικό κόστος είναι σημαντικό, παίζει ρόλο, θα πρέπει όμως να εξεταστεί το θέμα πιο ευρέως. Εγώ χάρηκα που είδα για αυτό, αυτή την πρόταση της μείωσης του 3% ότι είναι δυνατόν δηλαδή να βελτιωθούν οι, οι έλεγχοι χωρίς συμπληρωματικό κόστος και ήδη δυνατόν φαίνεται στα ιδιωτικά ταμεία να βελτιωθεί το ποσοστό σφάλματος κατά 3% χωρίς συμπληρωματικό κόστος. Αυτό είναι θαυμάσιο. Ίσως μπορεί να γίνει κάτι παρόμοιο και σε άλλους τομείς. Απλούστευση φυσικά λειτουργεί προς την κατεύθυνση αυτή. γιατί έτσι θα μπορούσαν οι κανόνες να είναι πιο αποτελεσματικοί, λιγότερο γραφειοκρατικοί και να μειωθεί έτσι το ποσοστό του σφάλματος χωρίς να αυξηθεί το κόστος. Τέλος, εδώ οδηγούμε αυτόματα στα συμπεράσματα, είναι σημαντικό να εξεταστεί το θέμα της αποτελεσματικότητας των σημερινών ελέγχων, γιατί έχουν την εντύπωση ότι αν δεν είναι ε, από υψηλή αποτελεσματικότητα ίσως χρειαστεί το αποδεκτό σφάλμα να οριστεί σε ένα επίπεδο που προϋποθέτει κάποια αποτελεσματικότητα. Από ό,τι κατάλαβα τον κύριο Καλάς δεν ισχύει αυτό. Αλλά υπάρχει ανάγκη να συνεχίσουμε να εξετάζουμε το στοιχείο αυτό για να δούμε ποιο είναι το κατάλληλο επίπεδο. Αυτέ είναι κάποιε από τι προσωπικέ μα σκέψει, όπω σα είπε κύριε Πρόεδρε γιατί το έγγραφο μα αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε προετοιμάσει. Εξετάζουμε ακόμα την ανακοίνωση τη Κομισιόν. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Σα ευχαριστούμε και για τι σκέψει που μα εκθέσατε. Ξέρουμε πόσο ευαίσθητο και σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Και γι' αυτό πρέπει να εκφράσουμε ευχαριστίες στο ελεγκτικό συνέδριο ότι αυτό το καυτό σίδερο το έθιξε, το άγγιξε στην τοποθέτησή του. Ζήτησε τον λόγο ο κύριος Καζάκα, συνάδελφος παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το επίπεδο πραγματικά αναβαθμισμένο υψηλής ποιότητας αυτού του εγγράφου που το διάβασα με μεγάλη προσοχή καθώς και το άλλο έγγραφο εργασίας το οποίο το συνοδεύει αυτό. Και επίσης ευχαριστούμε και για την εμβάθυνση, το βάθος των σκέψεων και προβληματισμών Υπάρχουν όμως εδώ διαφορετικά θέματα πράγματι που τίθενται. Πρώτα και κύρια, ακριβώς αυτό το οποίο αναφέρθηκε από το συνάδελφό μας ο Ντί πιο πριν. Επίσης και εγώ προσωπικά πιστεύω και σύμφωνα με αυτά τα οποία διάβασα για αυτό το θέμα και λαμβάνοντας υπόψη κυρίως επίσης αυτό που ο παλαιός μας συνάδελφος Χουάν Κολόνι Ναβάρ το δικαστήριο της Καταλωνίας ε, είχε αναφέρει και νομίζω ότι χρήσιμο θα είναι να έχουμε την υποστήριξη και παρακολούθηση των συναδέλφων και εκείνων που ε, μιλούν και ισπανικά και που μας δίνει μια πολύ αξιόλογη ε, παρουσίαση αυτής της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως θεωρώ ότι σύμφωνα με όσα γνωρίζω ο κύριος εισηγητής έχει δίκιο και αυτό είναι κάτι που ο ελεγκτής θα πρέπει πάντα να αποφασίζει και όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκείνη. Αληθεύει σίγουρα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την υπηρεσία εσωτερικών ελέγχων. Σίγουρα και η υπηρεσία εσωτερικών ελέγχων θα μπορούσε να τοποθετείται επ' αυτόν. Όμως τώρα από αυτά που διάβασα ως στοιχεία μέχρι τώρα πιστεύω ότι το ελεγκτικό συνέδριο δεν θα έπρεπε να ε, έχει ε, επ' απεμβολή να πεμπολεί ε, τις ευθύνες. Ένα άλλο θέμα και για την έκπληξη, για αυτό το 0,7% στο, στο, στο κόστος των διαρθρωτικών ταμείων. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορούσε να περιγράψει αναεπίπεδο την επίπτωση στο εθνικό, περιφερειακό, στο επίπεδο του ελεγκτικού συνεδρίου εσωτερικών ή εξωτερικών ελέγχων όλων αυτών ποσά που εκπλήσουν αυτά τα αριθμητικά μεγέθη. Θα πρέπει να δούμε ότι εδώ τριπλασιάζεται η προσπάθεια ελέγχου και αυτό ε, έχει τις επιπτώσεις του. Πέρα από αυτά τα δύο θέματα τα οποία αναφέρθηκαν, πιστεύω ότι υπάρχουν εδώ δύο σημεία πολύ σημαντικά που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ένα από αυτά είναι εκείνο που αφορά την διαφάνεια όλων των διεργασιών, όλης της διαδικασίας. Πιστεύω ότι άσχετα από τον ελεγκτή που θα πρέπει να λειτουργεί με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και αρχές, ότι θα πρέπει να είναι πραγματικά απαραίτητο και παραπάνω από χρήσιμο, απαραίτητο να μπορούμε να έχουμε άμεση επαφή με την πραγματικότητα και με τα σφάλματα τα οποία στην πραγματική ζωή σημειώνονται εδώ. Στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου γίνεται ένα βήμα προς τα εμπρός, διότι δίνονται παραδείγματα τα οποία καλά περιγράφονται και καλά εντοπίζονται, όμως δεν ταυτοποιούνται και δεν αναφέρεται ονομαστικά ποιος έχει κάνει αυτά τα λάθη και πού, σε ποια περιοχή, περιφέρεια ή ποια χώρα. Και γίνεται ένα βήμα εμπρό, δύο βήματα πίσω όμω. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να εκφράσω την θλίψη μου γι' αυτό. Θεωρώ απαραίτητο να γνωρίζουμε πολύ καλά γιατί πράγμα συζητάμε. Αν δεν γνωρίζουμε γιατί πράγμα κάνουμε λόγο και αν σε σχέση με τα σφάλματα τα οποία εδώ αναφέρονται, αν δεν γνωρίζουμε σε τι οφείλονται και ποιο τα προκαλεί, τότε χάνουμε τον έλεγχο και την ε, ε, εικόνα. Δεύτερο σημείο το οποίο θεωρώ ότι εδώ θεωρώ ότι δεν μπορώ να συμφωνήσω με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται σε αυτό το έγγραφο είναι το θέμα της απλούστευσης. Αναφέρει στη σελίδα 4 της ανακοίνωσης της ε, η Επιτροπή και το αναφέρω στα αγγλικά αυτό περίπλοκοι κανόνες και κριτήρια επιλεξιμότητας καμιά φορά είναι αναγκαία για να επιτευχθούν στοχοθετημένα αποτελέσματα πολιτικών που τα ωφελήματά τους ε, είναι χρήσιμα και όσον αφορά διεργασίες που μπορεί να υφίστανται κάποιο ποσοστό σφάλματος. Δηλαδή, αυτό σε σχέση με το θέμα για την απλούστευση στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν νομίζω ότι είναι η θετικότερη προσέγγιση για την επίλυση του προβλήματος. Πιστεύω ότι το μεγάλο πρόβλημα της απλούστευσης είναι ότι συνολικά οι νομοθέτες σε εθνικό επίπεδο, ευρωπαϊκό αλλά και περιφερειακό δεν λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις εκείνων που νομοθετούν. Όταν δηλαδή συγκεκριμένο κανόνα για επιλεξιμότητα υιοθετούν, δεν λαμβάνουν πάντα υπόψη το σφάλμα, το ποσοστό σφάλματος το οποίο μπορεί να ε, υπάρξει και που μπορεί να είναι και μεγάλο. Και εδώ έχουμε και το θέμα της διαφάνειας σίγουρα και είναι και το θέμα των συγκεκριμένων περιπτώσεων που απαιτείται διαφάνεια για αυτές. Και εδώ για την μηχανική αναζήτηση ε, του ποσοστού σφάλματος ε, πρέπει να του ποσοστού ανεκτού σφάλματος ε, είναι σημαντική η αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Αυτά τα δύο σημεία ήθελα να αναφέρω. Πρέπει να τα θεωρήσουμε ως απαραίτητα σημεία για τις συζητήσεις μας, για τις εργασίες μας και πέρα από αυτή την κοινοβουλευτική θητεία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την ωραία ανακοίνωση, την οποία περιμέναμε επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Νομίζω πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για το ότι την έχουμε τώρα αυτήν και το ότι με τα προβλήματα σε βάθος ε, τα φωτίζει και σε σχέση με την ε, ε, διατύπωση ανεκτός φάλμα σε μεγαλύτερο βάθος περνάμε είναι καλή λοιπόν αυτή η προσέγγιση. Στο τέλος τέλος ε, μια τέτοια συζήτηση και μια τέτοια απόφαση δεν θα μπορεί και δεν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη χωρί εμά και τη συμμετοχή μα. Θέλω να παρακαλέσω του συναδέλφου να διεξαγάγουμε τη συζήτηση τώρα για αυτά. Να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελληνικό Συνέδριο να συζητήσουμε αυτά τα θέματα σε βάθο με μεγάλη σοβαρότητα. Να δούμε πόσο αξιόπιστα είναι τα αριθμητικά μεγέθη επί των οποίων βασίζονται αυτά τα υπερδομήματα. Ε, ε, σε σχέση με τα, την, τις μαθηματικές ε, προσεγγίσεις ή υπολογισμούς, τι γνωρίζουμε για τα στοιχεία για τους ελέγχους από τα κράτη-μέλη. Πολύ λίγα. Από το 2006-2007 κάτι γνωρίζουμε. Αλλά έχουμε και κενά σχετικά με αυτά τα θέματα εδώ. Μέχρι το 2013 για τα επικαιροποιημένα προγράμματα με τη βάση με βάση αυτή τη ε, μέθοδο θα έπρεπε να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Έχω λοιπόν και σοβαρές αμφιβολίες για τα αριθμητικά μεγέθη των κρατών μελών. Έτσι όπως υποβάλλονται αυτά τα στοιχεία δεν υπάρχει δυνατότητα πια να δραστηριοποιηθούμε εμείς όπως πρέπει. Για κάτω από 1% δεν χρειάζεται να υπάρξει κάποια αντίδραση από πλευρά από πλευρά μα. Διερωτώ όμω, συμβαίνει πράγματι αυτό. Είναι δεδομένο αυτό και αξιόπιστο. Για την κατάσταση για τα διαθοτικά ταμεία βρίσκεται στα 3% και όχι στο 0,9%. Πρέπει να γνωρίζουμε λοιπόν πολλά περισσότερα για αυτά τα στοιχεία, τα αριθμητικά μεγέθη. Θέλω να ζητήσω το ελεγκτικό συνέδριο να ξαναεξετάσει αυτά τα στοιχεία. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να απαιτήσει κανεί προτού συνεχιστεί η συζήτηση για αυτά. Αυτό απαιτείται να γίνει. Να καλύψει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κενά. Το ανέφερε και ο επίτροπο Κάλλας. Τους τομείς που απουσιάζουν, που λείπουν ακόμα, τους χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Και με βάση τη νέα νομική βάση χρειαζόμαστε αυτά τα στοιχεία. Χρειαζόμαστε επίσης και τον πολιτισμό, κύριε Επίτροπε. Στην απαρίθμησή σας ο πολιτισμός δεν εντασσόταν στα στοιχεία που είχαν επισκοπηθεί. Και στην ερώτηση αυτή πόσο ο πολιτισμός δεν έχει συμπεριληφθεί, ίσω κάτι θα μπορούσατε να πείτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι οι τομείς που ασχολούνται με τη διαχείριση οι επιδοτήσεων να μπορούν να συμπεριλαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο και να εντάσσονται στην εξέταση από πλευρά μα. Να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι τομεί, αλλά και η ποιότητα των στοιχείων να αξιολογείται. Και νομίζω πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα των στοιχείων. Ο συνάδελφο Καζάκα το προανέφερε πιο πριν. Χρειαζόμαστε επίση με βάση αυτά τα στοιχεία ένα ranking, μια αξιολόγηση από πλευρά των κρατών μελών για να δούμε τι γίνεται και να δούμε και σε σχέση με τις περιφέρειες ranking, ιεράρχηση σφαλμάτων. Να δούμε πού βρίσκεται το πρόβλημα. Χτυπάμε με το πυροβόλο εναντίον όλων των στόχων, αλλά πρέπει να μπορούμε να διαφοροποιούμαστε, να ξέρουμε έναντι μιας περιφέρειας τι συμβαίνει, για να, να ε, γνωρίζουμε με βάση τα ελεγκτικά αυτά στοιχεία τι συμβαίνει επί τόπου. Στην ανακοίνωση δεν αναφέρονται πολλά για τον συσχετισμό κόστους και ελέγχου. Γίνονται κάποιες υποθέσεις που τις θεωρώ πολύ αμφισβητήσιμες. Σύμφωνα με αυτές τις υποθέσεις εργασίας, αυτές πρέπει να επανεξεταστούν. Όταν ε, ε, λαμβάνουμε κάποιες αποφάσεις δεν μπορούμε με βάση αυτά τα στοιχεία να αποφασίζουμε. Έκανε μια προσπάθεια να οικοδομήσει σε σαθρά θεμέλια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει όμως να είναι σταθερά και αξιόπιστα τα θεμέλια για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε. Με ενδιαφέρει λοιπόν πόσο έλεγχος, η ποιότητα ελέγχου αυτών των στοιχείων και το κόστος συναρτώνται. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν την ίδια ποιότητα στοιχείων και ελέγχων. Εκεί όπου έχει αμφιβολίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάρχουν ε, απαιτήσει να υπάρχουν ε, ε, κάποια διαφορετικά στοιχεία για τους ελέγχους, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία όμως αγνοούμε. Δεν τα έχουμε στη διάθεσή μας. Σημαντικό θα ήταν σε σχέση με τη συζήτηση να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση με βάση υποβολή βελτιωμένων ή αξιόπιστων στοιχείων. Και σίγουρα και από το Συμβούλιο θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε πώς αντέδρασε το Συμβούλιο σχετικά με όλα αυτά. Πρέπει να είναι αποφασισμένο το το, συμβούλιο, να, το Κοινοβούλιο να μπορέσει να διεξαγάγει αυτή τη συζήτηση ενωμένο εναντί ε, των ε, εταίρων του. Και πρέπει εδώ να τεθούμε στην πλευρά της ε, Επιτροπής για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Κύριος Ήτον παρακαλώ. Φαντάζομαι ότι μπορώ να πω ότι καλωσορίζω αυτή την προσέγγιση. Λυπάμαι και τον κύριο Κάλλας και τη διεύθυνσή του διότι από ό,τι ξέρουμε κάποιοι και εγώ, είναι ότι εμεί οι πολιτικοί είμαστε πολύ καλοί όταν θέλουμε να ξοδεύονται χρήματα για τα προγράμματα που ψηφίζουμε. Διότι τότε ίσω μα ψηφίσουν οι ψηφοφόροι, γιατί του δίνουμε χρήματα. Δεν θέλουμε περίπλοκε διαδικασίε που εμποδίζουν του ανθρώπου να αφαιρηθούν το πρόγραμμα. Δεν θέλουμε να ξοδεύονται πολλά για περίπλοκε διαδικασίε που ελέγχουν ότι ωφελούνται οι άνθρωποι τα χρήματα, διότι τα χρήματα θέλουμε να πηγαίνουν στα προγράμματα που ψηφίζουμε. Αλλά θα σας χυμίξουμε αν υπάρχει ένα πρόβλημα που βρίσκετε εσείς ή κάποιος άλλος. Ε, σφάλματα ή απάτες να διαπιστώνετε. Και δυστυχώς αυτή είναι η καποιος αλλος σφαλματα η απατες να διαπιστωνετε και δυστυχως αυτη ειναι η θεση που αντιμετωπίζετε. Στη δίκηση καμιά φορά ανησυχείτε για τους απλούς πολιτικούς στόχους που κρύβουν από πίσω περιπλοκότατα προγράμματα. Οι περισσότεροι παριστάμενοι στην αίθουσα το κατανοούν. Ξέρουμε ότι έλεγχος τρόπου δαπάνης των χρημάτων και σωστής χρήσης των χρημάτων δεν είναι τόσο διασκεδαστικό όσο το να δίνεις τα χρήματα εν πρώτης. Και το ελεκτικό συνέδριο εκεί πίσω έχει μεγάλο πρόβλημα, είναι πολύ καλή δική σας έλεγχη στην Κομισιόν. Βαρεμάρα, τι δουλειά να κάνουν αυτοί. Ο ελεγκτής θέλει να βρει πρόβλημα. Που σου ξέφυγαν εσένα. Και καλά τα καταφέρνει το συνέδριο. Εμείς, τώρα όχι εμείς, πάντα δύναμα απαλλαγή και άλλες χρονιές ανεξαρτήτως προβλημάτων. Θέλω Βρετανό πολιτικό. Εγώ που είμαι Βρετανός πολιτικός μάλλον, συγγνώμη. Θέλω μεγαλύτερη ειλικρίνεια. Όπως τα είπα ομά, χήμα και σταράτα στη δική μου μήνυ παρουσίαση. Ζήτησα στοιχεία για τα τελευταία χρόνια όπου μπορούμε εκεί να εκτιμήσουμε, να αξιολογήσουμε κατά πόσο οι διευθύνσει βελτιώνονται. πλησιάζουμε, τα καταφέρνουμε και εκτιμώ τη δουλειά που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δίνοντας κάποια στοιχεία, κάποια σημάδια για να κρίνουμε πώς πάει η δουλειά. Αν δεν έχουμε σωστά στοιχεία να κρίνουμε όμως, πάντα άνθρωποι σαν και εμένα θα σας ενοχλούν, διότι εκτίθενται και σα κυνηγάνε. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί στη συζήτηση. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι προσπαθείτε να κάνετε. Εγώ δεν είμαι πεπισμένο ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Δεν είμαι πεπισμένο για την ερμηνεία που θα δώσει Συμβούλιο και θα ήθελα πολύ να δω ποια είναι η άποψη του ελεκτικού συνεδρίου όταν καταλήξω κάποια άποψη. Βασικά, δώστε μας κάτι να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και να δουλέψουμε. Και περισσότεροι θα ευχαριστηθούν. Χρειαζόμαστε σωστά στοιχεία για αξιολόγηση, βαθμολόγηση, πολιτική εκτίμηση Γνωρίζετε πολύ καλά ότι θα σας παγιδεύσουμε κιόλα. Ε, Κύριε παρακαλώ. Yes, um, Μάλιστα. Ζεσταίνει την καρδιά του παλιού οικονομολόγου να δει κανεί το σημείο επαφή μεταξύ, ε, την εφαπτωμένη μεταξύ καμπύλη και ευθεία. Δύο προβλήματα βλέπω εγώ. Πρώτον, πρέπει να είναι δύσκολο να καθορίσει κανείς αριθμητικά στοιχεία σε μια καμπύλη για να ξέρει ποια είναι η μορφή της καμπύλης. Μπορούμε να ακολουθήσουμε την προσέγγιση που σχεγράφησε στην αρχή ο Επίτροπος ο κ. Κάλλας. Όταν λέμε αποδεκτό, ανεκτό επίπεδο, Υπάρχει και η θεωρία της εμπιστοσύνης στις κοινωνικές επιστήμες. Λες τους άλλους, θα τα καταφέρουμε, θα μειώσουμε τα σφάλματα, κίνδυνο απατών, τις απάτες που αξίζει να εξαλείψουμε. Τα υπόλοιπα τα αφήσουμε. Λέτε σε όλους τους άλλους λοιπόν ότι δεν θα το δούμε τα υπόλοιπα. Θα συνεχίσουμε Σκεφτήκατε πώς θα το προσεγγίσετε το θέμα. Μπορείτε να πείτε ότι πέραν αυτού θα κάνουμε και άλλους ελέγχους που ίσως σας εκπλήξουν και τελειώσει η καριέρα σας λέτε στους άλλους διότι διαφορετικά αν βλέμε στον κόσμο σε οποιοδήποτε σύστημα λέμε στον κόσμο ότι δεν μας νοιάζει αν κάνετε το ένα και το άλλο Εντάξει, εγκληματάκι είναι, αλλά εντάξει. Αυτό δημιουργεί κινδύνους. Το σκεφτήκατε, έχετε κάποιες ιδέες. Uh, uh, Συνάδελφοι, γνωρίζετε βέβαια κατά το παρελθόν το σύνολο της Επιτροπής όπως διαπιστώθηκε θεωρούσε αναγκαίο από αυτή την παγίδα στην οποία είχαμε βρεθεί να μην ε, ξαναπέσουμε, να πεγκλωβιστούμε αλλά και η επίπτωση και το λέω αυτό συνειδητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πολιτική για τις δαπάνες ακόμα πιο επιφυλακτική, η πιο δειλή κιόλα ακόμα μπορεί να πει κανείς έγινε και δεν μπορεί να είναι αυτό το νόημα, το εγχείρημα ενός προπολογισμού σε κάποιους τομείς ένας προϋπολογισμός λόγω μιας τέτοιας τάσης η επιφύλαξη σας το πω έτσι δεν μπορεί να δαπανηθεί σωστά και έχουμε τομείς πολιτικών και συμβαίνει αυτή, σε αυτή την ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με το κοινοβουλευτικό επίπεδο εμείς είμαστε πιο κοντά στους αρμόδιους από ό,τι άλλοι έχουμε πεδία πολιτικής όπου οι τίτλοι είναι και και κενά χωρίς ουσία. Όταν κάνουμε λόγο για παράδειγμα για τι γίνεται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καινή λόγοι είναι αυτοί. Άδεια και λύθη. Ε, και τότε σε σχέση με ένα ευρωπαϊκό τέτοιο πρόγραμμα Πώ μπορεί κανεί ε, σε σχέση με του κανόνε του παιχνιδιού να παροτρύνει κάποιον συμμετάσχει όταν η κατάσταση δεν ε, ενθαρρύνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να γίνεται λοιπόν αυτό. Το είχαμε στο παρελθόν και είχαμε δει αυτή την κατάσταση. Είχαμε σχεδόν δυσκολίε να εξηγήσουμε ότι ακριβώ μια επιτροπή ελέγχου προπολογισμών έχει θέσει ως έργο αυτό το θέμα ελέγχου και το αποδεκτό επίπεδο σφάλματος να το προσεγγίσει πιο αποτελεσματικά και καλύτερα. Γι' αυτό πρώτον είμαι ευγνώμων στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο όπου στην ανακοίνωσή του, του ε, αναφέρεται σε αυτό το καυτό πρόβλημα. Ήταν το πρώτο θεσμικό όργανο που το έκανε αυτό και μπορείτε πραγματικά να είστε υπερήφανοι γι' αυτό. Είναι επίτευγμα, δεν είναι απλό. Ήταν ένα σημαντικό επίτευγμα. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Κάλες, με όλα τα σημεία αυτά τα τα οποία αναφέρονται και έχουν προσθεθεί. Αυτά να ληφθούν με κάθε σοβαρότητα υπόψη. Και περάσατε τον Ρουβίκονα. Είναι απλό αυτό. Κάνατε ένα μεγάλο βήμα και έχετε ως κριτικούς εταίρους εμάς ε, με κριτικό πνεύμα στο πλευρό σας. Θέλουμε να γίνει καλύτερος ο προϋπολογισμός στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και κονδυλίων που διαθέτουμε. Και έχουμε και ένα επόμενο σημείο που πρόκειται στη συνέχεια για την το δεύτερο έγγραφο εργασίας ε, για την ε, αναθεώρηση ε, των δημοσιονομικών. Θέτουμε και αυτό το πρόβλημα, τίθεται αυτό το πρόβλημα με το ανεκτό επίπεδο σφάλματος ή κινδύνου και με τα βέλτιστα σημεία τα οποία αναφέρθηκαν από τον κύριο Μπονίτσι και από τον κύριο Λούντγκρεν και επίσης έχουμε άλλα θέματα όπως reputational risk, το θέμα δηλαδή κινδύνου στην αξιοπιστία, ή στο κύρος. Και εδώ πολιτικά πρέπει να δραστηριοποιηθούμε ως υπεύθυνοι για να είμαστε στο ορθό επίπεδο. Αλλά λαμβάνοντας υπόψη και την πραγματογνωμοσύνη βέβαια του ελεκτικού συνεδρίου, κάποτε πρέπει οι πολιτικά υπεύθυνοι, οι αιρετοί εκπρόσωποι να λαμβάνουν τις αναγκαίες αποφάσεις. Εδώ έχουμε κάποια παραδείγματα. Όταν κάποιες χιλιάδες ευρώ πέφτουν έξω για παράδειγμα όσον αφορά το επίδομα ε, ευρωβουλευτή για τους βοηθούς του ή κάποιος ε, επίτροπος ε, έχει κάνει κάποια πρόσθετα έξοδα σε σχέση με το, οικονομι... με το όχημα, υπηρεσιακό όχημα που του διαθέτουμε. Όμως εδώ πρέπει να δούμε την πραγματική διάσταση των κινδύνων. Από την άλλη πλευρά υπό το οικονομικό στοιχείο και στην διεθνή πολιτική και με τις ε, δαπάνες ε, που γίνονται από πλευράς μας ε, και τις δράσεις που υιοθετούνται να δούμε τις δυσκολίες που έγκυνται και όμως πολιτικά είναι πάρα πολύ σημαντικό παρότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος θέλουμε αυτά τα κονδύλια να δαπανώνται σε αυτές τις περιοχές έκδηλης κρίσης Πρέπει λοιπόν να χαιρετήσουμε αυτό το οποίο έγινε. Αναμένουμε λοιπόν την έκθεσή σας κύριε Μπονίτσι από πλευρά σας, από δεν πρέπει να πεμπολίσετε αυτό το θέμα, πρέπει να δοθεί συνέχεια και να το παρακολουθήσουμε. Από κοινού, εμείς οι τρεις που το παρακολουθούσαμε, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωβουλή, πρέπει να επιμείνουμε ο τέταρτος παίκτη, το Συμβούλιο, να αναλάβει τις ευθύνες του και να πει ποιε είναι οι πεπιθήσεις του. Δεν το έκανε μέχρι τώρα το Συμβούλιο και είμαι ευγνώμων για αυτά που είπε η κυρία Γκρέσλε, τα σχόλιά της και μπορεί και να μας βοηθήσει το ελεκτικό συνέδριο και να μπορούν να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Αυτά τα αριθμητικά μεγέθη τα οποία χρειάζονται να δοθούν σε σχέση με τα στοιχεία που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ξανασχοληθούμε με αυτά, να τα ξαναδούμε. Διότι αν αυτό θα ήταν το μήνυμα το οποίο περνάει με 0,7 ή 0,8% σφάλμα όλο και όλο, ε τότε συγγνώμη δεν θα υπάρχει καμιά δικαιολογία πια ακόμα και για τα κράτη-μέλη που μας λένε ότι συντρίβονται από τις δαπάνες και από τις προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν για τα διαθωτικά ταμεία για παράδειγμα. Και μετά όταν έχουμε το 11% το οποίο διαπιστώνεται από το ελεγκτικό συνέδριο, τι γίνεται και μετά παίρνει κανείς μια τελείως διαφορετική γεύση και επίγευση και βλέπει ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να, να υπάρξει πρόοδος σε σχέση με αυτά τα στοιχεία. Έχει απόλυτο δίκιο η κυρία Γκρέσλε. Αυτά είναι τα ουσιοδέστερα στοιχεία. Και φυσικά θα θέλαμε να εξειδικεύσουμε περισσότερο τα πράγματα. Αν θα κινητοποιηθούμε προς την κατεύθυνση των περιφερειών ή προ τα κράτη-μέλη. Εδώ είναι καυτό το θέμα αυτό και αξίζει να το ξαναδούμε, να το ξαναεξετάσουμε και συγκεκριμένα να το αντιμετωπίσουμε για να επιτευχθεί πραγματικά επίπεδο αξιόπιστο αυτό το στοιχείο. Τι γίνεται με την ποιότητα των κρατών μελών. Θα ήταν θαύμα αν υπήρχε το ίδιο επίπεδο ε, ποιότητας που διασφαλίζεται από κοινού από όλα τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, Έχουμε κάποιους μήνες μπροστά μας ακόμα, έχουμε κάποιο χρόνο, πρέπει να δραχθούμε τις ευκαιρίες να χρησιμοποιήσουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Αναζωογονήθηκε η συζήτηση. Σας ευχαριστούμε λοιπόν θερμά, πιστεύω εγώ, αυτό πρέπει να πούμε με κάθε μετριοφροσύνη. Σας ευχαριστούμε για τις πρόοδους που επετέχθησαν. Και εμεί ω ε, Επιτροπή ε, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου το προπολογισμό, θα δώσουμε συνέχεια. Θα παραμείνουμε στο παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα, δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος, ε, κύριε Κάλλα, κύριε, κύριε Μπονίτσι, θέλετε να κάνετε κάποιε παρατηρήσει. Ο κύριο Κάλλα, λοιπόν, παρακαλώ. Μικρέ παρατηρήσει. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σα. Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι είμαστε σύμμαχοι. Εγώ δεν παραπονέθηκα ποτέ για τη συνεργασία μεταξύ τη Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια τη θητεία μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλή συνεργασία και με το ελεκτικό συνέδριο. Σχόλια. Πάνω σε αυτά πήγε ο Ήτον Χάρης. Ότι θα δημιουργήσουμε σύστημα βαθμονόμησης. Benchmarking και όπως είπατε είναι επίμαχο ζήτημα. Μερικοί πολιτικοί και μερικοί εκπρόσωποι της κοινή γνώμης δεν θέλουν τη βαθμονόμηση γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να γενικολογεί κανείς. Αλλά μέσω συστήματος βαθμονόμησης θυμόμαστε πάντα ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. και ο καλύτερος αριθμός είναι οι λεπτομέρειες, όπου εκεί μπορεί να βρεις διάφορους διαβόλους διαφόρων μεγεθών για το βέλτιστον. Δεν το βρίσκουμε μέσα του οικονομικού μοντέλου μόνο, έχουμε βρει το 4% και τα διαθετικά ταμεία, ίσως να είναι 5%. Ανάπτυξη της υπαίθρου μικραίνει, από, μειώνεται από 8% στα 5%. Η ε, κυρία Γκρέσλερ έθεσε το ερώτημα για άλλους τομείς. Πήραμε τους πρώτους τομείς εμείς. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά για να προχωρήσουμε και βέβαια υπάρχει και σχετικό πρόγραμμα να καλύψουμε και τους άλλους τομείς. Μπορώ να πω μόνο ότι έχει κάποια απόχρωση έννοια του διοικητικού κόστους. Μπορούμε να μειώσουμε το επίπεδο ανεκτού κινδύνου. Αλλά το κόστος του ελέγχου στο διοικητικό τομέα είναι αρκετά υψηλό. Δεν ξέρω το ακριβές ποσό, αλλά υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος για σφάλματα σε αυτόν τον τομέα από ότι σε άλλους τομείς και δημιουργείται και κίνδυνος για τη φήμη, το reputation risk. Άρα είναι και άλλες στοιχείες που ληφθούν υπόψη πέραν του βελτίστου οικονομικού. Ο κ. Μπέρς και η κυρία Γκρέσλερ αναφέθηκαν σε κάτι στην αξιοπιστία των στοιχείων. Βεβαίως έχουμε διορθώσει τα στοιχεία για τα οποία είχαμε υπόνοιες ότι δεν είναι σωστά. Ας συμφωνήσουμε όμως επί της μεθόδου. Α συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο, με το Κοινοβούλιο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ας συμφωνήσουμε όλοι μαζί και με το Ελεκτικό Συνέδριο τη μέθοδο. Και μετά ρυθμίζουμε τα στοιχεία. Τεράστιο έργο μας περιμένει αν θέλουμε να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο. Το ευαίσθητο θέμα είναι ποιος καθορίζει εν τέλει τα στοιχεία και τον ανεκτό κίνδυνο. Πέραν του οικονομικού βελτίστου αριθμητικού στοιχείου. Μία άποψη είναι ότι ελεγκτής το καθορίζει. Άλλος ότι οι νομοθέτες πρέπει να αποφασίσουν. Βεβαίω, ο ελεγχόμενο είναι ο τελευταίο που θα το προτείνει αυτό. Μπορούμε να προτείνουμε τρόπου υπολογισμού αλλά η απόφαση πρέπει να είναι διοργανική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σαφή υποστήριξη που έχετε, μας δώσατε ότι χρειάζεται σαφέστερη περιγραφή των θεμάτων περί απαλλαγής και έλεγχου. Προσβλέπω σε συνέχιση των προσπαθειών. Επί σειρά ετών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε συζητήσει τους διαβόλους των λεπτομεριών και σε ποια αποτελέσματα πρέπει να καταλήξουμε μέσω οποίων υπολογισμών. Εγώ είμαι ενθουσιώδης. Ε, χαίρομαι όλους ιδιαίτερα που διεξήχθη αυτή η συζήτηση και σας ευχαριστώ. Από πλευρά ελεκτικού συνεδρίου υπάρχει κάτι με την... Ε, θα θέλαμε να περιμένουμε να υπάρξει αυτή η γνωμοδότηση. Σας το είπα πιο πριν. Ναι, όπως σας είπα, το ελεκτικό συνέδριο συζητά την ανακοίνωση να πω ότι είναι πολύ καλή αυτή η εξέλιξη. Δηλαδή το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοίμασε ένα έγγραφο, το οποίο έγγραφο προσπαθεί αντικειμενικά να βρει λύση για κάποια σημεία. Είχα προαναφέρει ότι δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεώθηκε να περιοριστεί λόγω των διαθεσίμων πληροφοριών. Ίσως αυτό που πρέπει να γίνει είναι να κατά πόσο αυτή η βάση δεδομένων μπορεί να βελτιωθεί. Δεν είναι θέμα δικό μας να ελέγξουμε τις πληροφορίες, αλλά πρέπει να είναι στιβαρές αυτές οι πληροφορίες για να είναι σωστή η ζωή στη συζήτηση. Και δυστυχώς πρέπει να γίνει και άλλη δουλειά από τον γνωστό ύποπτο. Χαίρομαι για τη συζήτηση. Το θέμα του ανεκτού ποσοστού κινδύνου είναι κάτι που πλανάται επί σειρά ετών και εν τέλει βλέπουμε κάτι που μας δίνει και άλλες πληροφορίες που δεν υπήρχαν. Και οι πληροφορίες αυτές μας επιτρέπουν τη διεξαγωγή μια μελλοντική επικοδομητικής συζητήσεως. Αυτά και ευχαριστώ. Πολύ ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα. Προφταίνουμε να εξετάσουμε το τελευταίο σημείο. Σημείο πέντε 5 στην ημερήσια διάταξη. Θα ήταν καλό αν έμεινε εδώ ο κ. Αντιπρόεδρος, γιατί και εδώ παίζει ένα ρόλο το ανοιχτό επίπεδο κινδύνου για να το δω αυτό. Σημείο 5. Ενδιάμεση επελεξάρση του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013. Μπορούμε νομίζω να το εξετάσουμε σχετικά γλίγορα. Υπάρχουν δύο έγγραφα εργασία για το θέμα αυτό. Όπως ξέρετε έχουν ήδη παρουσιαστεί στο παρελθόν τα έγγραφα αυτά. Ähm, Sie haben das... Äh, η αρμόδια βέβαια είναι η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Αυτό είναι σημαντικό για μας ως Επιτροπή Ελέγχου του Ξέρετε ότι υπήρχαν ορισμένοι που αναρωτιόντουσαν ποια είναι η σχέση μας ακριβώς με το προπολογισμό, αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε να παίξουμε ένα συγκεκριμένο ρόλο το βλέπετε ότι το έχουμε συνοψίσει σε λίγα κεντρικά θέματα που ελπίζουμε να γίνουν δεκτά από την επισουσία αρμόδια Επιτροπή ε, το θέμα του ενεκτού σφάλματος. Το χαιρετίζουμε και καλούμε την Κομισιό να υποβάλει κάποιες προτάσεις. Σήμερα νομίζω προχωρήσαμε. Σημειώνουμε επίσης και είμαστε και ιδιαίτερα είμαστε εδώ για, προς το ηλεκτρικό συνέδριο. Θα πρέπει δηλαδή να σκεφτούμε στο μέλλον εάν μια πολιτική δεν πετυχαίνει του στόχου της, με την πάροδο πολλών ετών θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια μαζική μεταρρύθμιση ή μάλιστα να επανεξετάσουμε ίσως να καταργήσουμε αυτή την πολιτική. Στη γνωμοδότησή μας τονίζουμε το θέμα των εθνικών διοικητικών δηλώσεων για να μπορέσει έτσι να ενδυναμωθεί η υποχρέωση λογοδοσίας των κρατών μελών. και νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε αφορά την καθορισμένη διαχείριση των πόρων μόνο αν έχουμε ένα είδος κοινοτική έγκρισης για τις υπηρεσίες εκείνες των κρατών μελών που διαχειρίζονται τα χρήματα αυτά. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά σημεία νομίζω που παίζουν εδώ ένα ρόλο. Ελπίζουμε ότι η Επιτροπή Προπολισμών θα δεχθεί αυτά τα σημεία. Θα με ενδιαφέρει να ακούσω τις αντιδράσεις σας από αυτού. Υπάρχουν τροπολογίες. Äh, ναι, η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών προβλέπεται για το μεσημέρι της 27ης Ιανουαρίου. Ποιος θα θέλει το λόγο παρακαλώ. Κανένας δεν θέλει. Α, όχι. Ο κύριος Γκρέι, παρακαλώ κύριε Γκρέι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ναι. δεν ήθελα να πω δύο λόγια για τις πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες που έχετε εδώ υποβάλει. Γιατί προφανώς ε, για την ενδιάμεση επανεξάρτηση ε, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία. Οι παρατηρήσεις σας ζητούν παραδείγματος χάρη μια ε, ισορροπία μεταξύ των οικονομικών ε, ε, ελέγχων και των ελέγχων της διαχείρισης. εκεί υπάρχει αυτή η έννοια της μοιρασμένης διαχείρισης και γι' αυτό εμείς ήδη κάνουμε αυτό που ζητάτε και επενδύουμε πολλά σε αυτά. Τώρα, έλεγχη απόδοση, Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι θέλετε. Για όλους τους τομεί πολιτική, βέβαια έχουμε μια αξιολόγηση, ενδιάμεση αξιολόγηση εκ των υστέρων αξιολόγηση και συγκρίνουμε τα αποτελέσματα με αυτό που είχαμε κατά νου αρχικά. Υπάρχουν λοιπόν οι σωστοί μηχανισμοί αξιολόγησης υποχρεωτικά μέσα στα πλαίσια του δημοσιονομικού κανονισμού. Προτείνεται επίσης η Κομισιόν να αξιολογεί και να πιστοποιεί αν θέλετε τις εθνικές υπηρεσίες. Αυτό γίνεται για έμεση διαχείριση αλλά για μοιρασμένη διαχείριση ίσως θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη η διαδικασία και θα καθυστερούσε την εφαρμογή του προγράμματος εάν η Κομισιόν πρόκειται να πιστοποιήσει αυτές τις υπηρεσίες. Αυτό που κάνουμε είναι ότι καλούμε τα κράτη-μέλη να ε, πιστοποιήσουν τις υπηρεσίες και εμείς ελέγχουμε το έργο που έχουν επιτελέσει τα κράτη-μέλη. Και μετά μπορεί ίσως να χρειαστεί να βελτιωθεί το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε. για τι εθνικέ δηλώσει, συζήτηση που κάνουμε έχουμε το άρθρο 53 του δημοσιονομικού κανονισμού που προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι το τηρούν τα κράτη-μέλη και για μια χώρα που δεν το τηρούσε κινήσαμε διαδικασία παραβάση. Άρα κράτη-μέλη προχωράνε πιο, πιο πέρα από τις απαιτήσει του άρθρου 53 Τις υποστηρίζουμε εμείς αυτές και βελτιώσαμε και τις κατευθύνες γραμμές για τα ερωτικά ταμεία για να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός αυτό. Κάτω χώρε, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία και Σουηδία παραδείγματος Χάριν. χρειάστηκαν κάποια βοήθεια για το πώς θα πρέπει να διατυπώσουν τις εθνικές αυτές δηλώσεις. Στο σημείο 4 λέτε ότι για ορισμένε ε, πολιτικές δεν μπορεί να υπάρχει πλήρη λογοδοσία και θα πρέπει να τροποποιηθούν οι διαδικασίες στην περίπτωση αυτή. Ναι, αυτό είναι κάτι που λαμβάνει υπόψη στην Κομισιό. Πολλές φορέ έχουμε καταλή... ε, καταργήσει κάποιε διαδικασίε γιατί θεωρούσαμε ότι δεν απέδαν το αποτέλεσμα. Παραδείγματο χάρη είναι, έχουμε εδώ το παράδειγμα των ενισχύσεων για, ε, για το Λίνο. Ή έχουμε τον κανονισμό 2013 που βολτιώνει κάποιες πολιτικές για να μπορέσει να βελτιωθεί η λογοδεσία. Ο κύριο Φίγκαλ προηγουμένως εξήγησε τι γίνεται στον τομέα της εκπαίδευσης κλπ. Το ανεκτός κίνδυνο συζητήθηκε ήδη. Αυτά είναι κάποια πρώτα σχόλια που έχουμε για τις ιδέες που έχετε παρουσιάσει εδώ. Ευχαριστώ. Πρώτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιος άλλο που έχει κάποια παρατήρηση, όχι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, επαναλαμβάνω, η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι 12 το μεσημέρι της 27 Ιανουαρίου. Πέρασε του σημείου αυτού και πέρα στις ημερησίες διάταξης ε, για σήμερα, γιατί όπως είπαμε η συζήτηση για την έκθεση Δεμπλάτια θα γίνει το Φεβρουάριο. Δεν θέλω να σας υπενθυμίσω, ιδίω ο προσώπης των πολιτικών ομάδων, ότι αύριο θα αρχίσουμε στις 9 με δύο ψηφοφορίες. Στις 9 ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποτελεσματική και πολύ καλή συνεργασία σήμερα το απόγευμα. Ελπίζω να συνεχίσουμε το χρόνο πέρασε συνεδρίαση μέχρι αύτο το πρωί 9.